Παρακαλώ, θα ήθελα να καθίσετε για να ξεκινήσουμε. Θα συνεχίσω στην Ιταλική γλώσσα. Επαναλαμβάνω, θα συνεχίσω στην Ιταλική γλώσσα, λέει η Πρόεδρος απειλώντας. Έχουμε μαζί μας την Υπουργό Πολιτισμού της Λετωνίας. In Italian. Allora, eh, intanto, buon Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους. Θέλω να σας ευχηθώ, να μου επιτρέψετε να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλή δουλειά, τις θερμότερες ευχές μου και στην Υπουργό της Λετωνίας, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία ήλθε να μας επισκεφτεί και η οποία θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας της. Πριν ξεκινήσω όμως την συνάντηση αυτή, τη συνεδρίαση αυτή, πριν αναφερθώ στην ημερήσια διάταξη, όπως είχαμε ήδη προβλέψει, νομίζω ότι θα ήταν σωστό, λόγω των αξιών με τις οποίες ασχολείται η Επιτροπή μας, να κρατήσουμε ενός λεπτού ε, σιγή προς, στιγμή, προς τιμήν των θυμάτων που ιδιαίτερα στην Γαλλία ήταν πάρα πολλά θύματα, σκοτώθηκαν με βάρβαρο τρόπο και οι δημοσιογράφοι του Σαρλί και οι πελάτες του καταστήματος Κοσέρ και οι δύο αστυνομικοί, οι δύο νέοι αστυνομικοί και τόσα θύματα επίσης στην Ιγυρία τις τελευταίες μέρες και στον Ήγυρα. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε αυτά. Νομίζω ότι πέρα από το, ε, ένα λεπτό σιγή το οποίο τηρήσαμε στο Στρασβούργο θα πρέπει και εδώ εμείς σαν Επιτροπή που είμαστε υπέρ της ελευθερίας της πολιτισμικής και υπέρ της ελευθερίας του τύπου να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, <clears throat> να πω ότι εξετίμησα δεόντως το ότι η υπουργό ανέλαβε την πρωτοβουλία τις τελευταίες ημέρες να προτείνει μια κοινή δήλωση όλων των Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κοινή δήλωση η οποία να καταδικάζει αυτές ε, τις ενέργειες και να υπογραμμίζει ότι πάντα προασπίζουμε τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, για το σημείο 5 πιο ειδικά, να θυμίσω ότι αφορά στην Λετωνική Προεδρία, κυρίως μέσω της έκθεσης της κυρίας Ντιμπάτσκα, για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια μέσω γραπτής πρωτοβουλίας. Είναι κάτι το οποίο ε, είναι στην ίδια φάση, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, ε, με το πρόγραμμα ε, Juncker για την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη λοιπόν θα ασχοληθούμε με το θέμα των επενδύσεων του τύπου και η πρωτοβουλία της Μπολόνια είναι μια καλή πρωτοβουλία και θα πρέπει να προχωρήσουμε και να δούμε πού βρισκόμαστε το ταχύτερο δυνατόν. Λοιπόν, πάντως ελπίζω να συμφωνείτε με αυτή τη μικρή τροποποίηση. Συνεχίζουμε. Έρχομαι στα πρακτικά της 1ης και της 2ης Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσεις, αλλιώς θα θεωρηθούν δεκτέ. Και να σας δώσω κάποιες επιπλέον πληροφορίες τώρα και γύρω από τις δυνατότητες διερμηνίας σε όλες σχεδόν τις γλώσσες. ρούμένο e, e, anche eh, in και φυσικά αντί για λιθουανικά έχουμε λετονικά για ευνόητους λόγους. Να σας ενημερώσω επίσης και σε σχέση με τη συμμετοχή μας στο νέο δίκτυο mainstreaming για την ισότητα των ευκαιριών στην οποία συμμετέχουν όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πρόθεση αυτής της ομάδας είναι να εργαστεί σε στενή συνεργασία με τις, με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θα πρέπει όλοι οι εισηγητές να λαμβάνουν υπόψη την διάσταση αυτή της ισότητας των ευκαιριών. Θα υπάρξει στενή συνεργασία και με την Επιτροπή Γυναικών και σε σχέση με τις εκθέσεις της Επιτροπής αυτής και με τις πρωτοβουλίες γενικότερα της κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής. Για το σημείο 4, φτάσαμε λοιπόν στο σημείο 4, είναι το βασικό ε, σημείο της παρουσίασής μας σήμερα. Θα ακούσουμε τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας και αυτό θα ακολουθηθεί από μια ανταλλαγή απόψεων την οποία θα έχουμε με την Υπουργό. Σας καλωσορίζω για μια ακόμη φορά, Υπουργέ. Γνωρίζετε ποια είναι η μέθοδος την οποία θα ακολουθήσουμε. Μετά από εσά θα πάρει το λόγο άλλωστε και η υπουργό Εκπαίδευσης της Λετωνίας, η οποία είναι ήδη παρούσα και θα μπορέσει να κάνει και αυτή την παρέμβασή της. Θα ακούσουμε λοιπόν μέσα σε 15 λεπτά τις προτεραιότητές σας και μετά θα πάρουν τον λόγο οι συνάδελφοι για να θέσουν εφόσον το επιθυμούν ερωτήσεις και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις μέσα σε 30 περίπου λεπτά. Θα κάνουμε δύο σειρές ερωτήσεων Αλλιώς θα δούμε μήπως χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος. Τώρα δίνω αμέσως το λόγο λοιπόν στην Υπουργό λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε μια στρατηγική συγκυρία. Ξεκινάει ουσιαστικά η κοινοβουλευτική περίοδος, Συναντηθήκαμε ήδη με την αρμόδια επίτροπο, θα συναντηθούμε και με τον επίτροπο Έτιγκερ σύντομα στο τέλος του μήνα και θα στείλουμε νομίζω, θα λάβουμε μάλλον ένα ισχυρό μήνυμα από πλευράς της Προεδρίας για να υπάρξει μια μεγαλύτερη προσήλωση στα θέματα του πολιτισμού και στα θέματα της παιδείας, στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης και το θέμα του πολιτισμού και τις σχέσεις της με την οικονομία και την ψηφιακή κυρίως οικονομία. Αυτές είναι οι προθέσεις μας για τους επόμενους μήνες. Έχετε το λόγο Υπουργέ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από πλευράς μου θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ ώστε να συζητήσω με την Επιτροπή σας για πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα και που έχω και την ευκαιρία να ακούσω εσάς, τις ιδέες σας, τις ανησυχίες σας, ε, τις προτάσεις σας. Ε, για να σεβαστώ και τη γλωσσική ε, πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα, τη λετωνική. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, για άλλη μια φορά θέλω να εκφράσω την τιμή που νιώθω που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες ε, της ε, Λετωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτισμού και της παιδείας ε, μετά από την πολύ επιτυχή Ιταλική Προεδρία. Πρώτα απ' όλα από πλευρά μου θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και την υποστήριξή μου στη Γαλλία και το λαό της μετά από την τραγωδία στο περιοδικό Σαλίεμπτο το ένα λεπτό που τηρήσαμε προλίγου για να φόρο φοροτιμήσεις στους ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους, ε, στους δημοσιογράφους, στο προσωπικό. Όλο αυτό μας υπενθυμίζει ότι είμαστε υπέρ των ενωμένων αξιών της Ευρώπης. που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία. Οι υπουργοί πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωση ανέλαβαν δράση πολύ γρήγορα και αυτό με συγκινεί. Υποστήριξαν την πρωτοβουλία που εγώ και ο υπουργό πολιτισμού της Γαλλίας ε, ξεκινήσαμε με μια ανακοίνωση καταδικάση αυτής της βαρβαρή ενέργειας. Και όλοι οι υπουργοί εξέφρασαν το ότι η ελευθερία των τεχνών και της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ. Και αυτό δείχνει ότι μπορούμε να βασιστούμε ένα στον άλλο σε τόσο δύσκολε εποχές. Μια τέτοια αρχή προεδρία μας διδάσκει πολλά. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε για να ενισχύσουμε και να προωθήσουμε την κατανόηση των κοινών μας αξιών. Πρέπει να συνεργαστούμε ώστε έξυπνα και σοφά να δημιουργήσουμε ένα ζωτικό χώρο όπου οι διάφοροι πολιτισμοί και οι διάφορες νοοτροπίες ε, δεν θα χωρίζουν την κοινωνία αλλά θα αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο την πρόωθηση επικοδομητικών συζητήσεων και σύσταση μιας εναρμονισμένης κοινωνίας. Τα όσα έγιναν στο Παρίσι έδειξαν ότι στον κόσμο μας ε, τα, οι διενέξεις γίνονται πιο οξύες μεταξύ διαφορετικών αξιών και απόψεων. Εδώ λαμβάνει περισσότερη αξία λοιπόν ο πολιτισμός. Δεν είναι απλά κάτι που απαντάμε καθημερινά στη ζωή μας σε μουσεία και σε άλλα σημεία. Ο πολιτισμός ε, είναι κάτι βαθύτερο. Εκφράζει διάφορες απόψεις και τρόπους συμβίωσης. Ο Ιμαν Ζήντος, ε, λετωνός είπε ότι ο πολιτισμός αποτελεί τη συνείδηση ενός έθνους. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό καθήκον να συνεργαστούμε ώστε οι διαφορετικοί λαοί και χώρες μας να ζήσουν σε αρμονία με τις νοοτροπίες τους και με τη συνείδησή τους. Αξιότιμα μέλη, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, έχοντας όλα αυτά στο μου θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις ε, λετονικές προτεραιότητες ε, στον τομέα του πολιτισμού. Ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ε, είναι πλέον πολύ σημαντικό κομμάτι της ε, πολιτικής ε, στην Ευρώπη. Λόγω της αποδεδειγμένης ικανότητας του τομέα να εξασφαλίσει έξυπνη, βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη και να βελτιώσει την ενιαία ψηφιακή αγορά. Η δημιουργικότητα που αποτελεί το βασικό πόρο των δημιουργικών ε, βιομηχανιών είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο του πολιτισμού αλλά και άλλων τομέων. Έχουμε γνωστά παραδείγματα, για παράδειγμα την ψηφιακή οικονομία, τον τουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων και δημιουργική σκέψη στη διάρκεια της παιδείας, τις νέες πολιτιστικές υποδομές ε, στα διάφορα εδάφη μας ε, και μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Νοέμβριο πέρυσι το Συμβούλιο συζήτησε τη συμβολή του πολιτισμού και των δημιουργικών ε, κλάδων ε, στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Ε, Το Συμβούλιο επικεντρώθηκε στη σπουδαιότητα αυτών των κλάδων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπό τη μορφή crossover όπως ονομάζεται στα αγγλικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ο όρο. Κύριε Προτεραιότητα τη Λετωνική Προεδρία είναι να συνεχίσει να ενισχύει την κατανόηση των υπευθύνων χάραξη πολιτική για τη θετική επιρροή του πολιτισμού στην κοινωνία μα, ώστε να βρει νέε λύσει και να διασφαλίσουν την αηφορία και τη βιωσιμότητα τη κοινωνία και τη οικονομία, χωρί αποκλεισμού. Η Λετωνική Προεδρία θα βασιστεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διασταύρωση, το crossover αυτό μεταξύ του πολιτισμού και των δημιουργικών κλάδων. Έχει έρθει η στιγμή για να το συζητήσουμε όλα αυτά ευρέω σε διάφορα φόρα, διότι η συμβολή του πολιτισμού και των λοιπών κλάδων είναι πλέον αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα θέλαμε όλοι μας να εστιαστούμε στη σπουδαιότητα των εθνικών και περιφερειακών παραγόντων για να προωθήσουμε αυτές τις πολιτικές. Θα θελήσουμε τα συμπεράσματα αυτά του Συμβουλίου να υιοθετηθούν στο Συμβούλιο του Μαΐου φέτος για να επεκτείνουμε τις συζητήσεις που έχουν γίνει στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσουμε δύο διασκέψεις της Προεδρίας στη Ρήγα από τις 11 μέχρι τις 13 Μαρτίου. Αυτές οι διεθνείς διασκέψεις θα λάβουν χώρα την ίδια εποχή με την ετήσια εβδομάδα δημιουργικότητας ε, στη Λετωνία, στη Ρήγα, που οργανώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ώστε να ενισχύουμε τον πολιτισμό και άλλες πολιτικές, όπως για παράδειγμα την οικονομική και περιφερειακή πολιτική. Μια τέτοια προσέγγιση εδώ και πολλά χρόνια μας προσφέρει μια σταθερή βάση για προώθηση της συνεργασίας ε, και της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορών κλάδων. Είστε λοιπόν προσκεκλημένοι να συμμετάσχετε σε αυτές τις διασκέψεις. Μπορείτε ελεύθερα να εγγραφείτε για αυτές, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ε, φυσικά εφόσον τηρήσετε τις προθεσμίες. Σκοπός της διάσκεψης είναι να εστιαστούμε στα κυριότερα παραδείγματα μεταξύ δημιουργικής συνεργασίας και πολιτισμού και να βρούμε τρόπους ενίσχυσης αυτής της συνεργασίας. Η δεύτερη διάσκεψη θα αφορά μια συζήτηση σε βάθος σε σχέση με την αλληλεπίδραση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του design και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ώστε να προσεγγίσουμε αυτά τα τρία στοιχεία, δημιουργώντας ένα ζωτικό χώρο υψηλής ποιότητας ε, για τους λαούς μας, τόσο για την εργασία όσο και για τη διαβίωση. Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμβολή της Επιτροπής σας στην πρόθεση της ανάπτυξης του πολιτισμού και της δημιουργικής πολιτικής Θέλω να εκφράσω την επιθυμία μου να συνεργαστούμε μαζί ώστε να συνεργαστούμε με τους υπευθύνους χαράξης πολιτικής στον τομέα αυτό. Αξιότιμα μέλη, η άνοιξη του 2015 θα υπάρξει εξαιρετικά σημαντική. Αναμένουμε μεσοπροθεσμία αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Στα τέλη του 2014, η, η Υπουργοί Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνάντηση του Συμβουλίου συζήτησαν για τη συμβολή του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας ε, στους στόχους της στρατηγικής 2020 και τόνισαν τρία πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Πρώτα απ' όλα ο πολιτισμός και η δημιουργική κλάδη αποτελούν ε, την ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης. Ε, δεύτερον, το δυναμικό αυτών των κλάδων πρέπει να είναι ελκυστικό, υψηλής ποιότητας ε, και πολιτιστικού περιεχομένου. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Τρίτον, ο πολιτισμός αποτελεί αξία από μόνος του. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας μοναδικός πόρος έμπνευσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας που συμβαδίζει με την εθνική μας και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αποτελεί σημάδι που χαρακτηρίζει την ταυτότητά μας ε, και τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν να στείλουμε και εμείς και να προωθήσουμε αυτά τα μηνύματα ώστε να βεβαιωθούμε ότι η συμβολή της δημιουργικότητας και του πολιτισμού θα αποτελέσει γεγονός ε, για την ε, έξυπνη ανάπτυξη της Ευρώπης και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να σας προσθέσω τώρα τις ε, προτεραιότητες για την οπτικοακουστική πολιτική. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ είπε ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν έχει αποφασίσει ότι η κεντρική πτυχή αυτής της πολιτικής θα είναι οι καταναλωτές της αγοράς με τις ηλεκτρονικές τους συσκευές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, μουσική και ταινίες από οπουδήποτε στην Ευρώπη. Δεδομένου αυτού η Κομισιόν ανέλαβε να υποστηρίξει την ανάπτυξη του πολιτισμού και των ε, δημιουργικών κλάδων και τους παραγωγούς περιεχομένου, τα ευρωπαϊκά μέσα και να αναπτύξει τον κανονισμό για το copyright. Η Κομισιόν επίσης τόνισε τη σπουδαιότητα της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ως ε, Λετωνή υπουργό Αρμόδια για τους τομείς αυτούς, ε, συγχαίρω την Κομισιόν για αυτές τις δηλώσεις της. Ε, θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται με τέτοιο τρόπο η σπουδαιότητα του πολιτισμού και του δημιουργικού τομέα. Βάση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών είναι η ελευθερία, η πολυμορφία, και η διαφορετικότητα των πολιτισμών που εκφράζονται μέσα στο περιεχόμενο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο που θα διατίθεται στους ε, πολίτες μας θα είναι υψηλής ποιότητας, πολυμορφικό ε, και θα ε, στηρίζει τις αξίες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η νέα γεωπολιτική κατάσταση και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός οδηγούν σε μια νέα ανάγκη επανασχεδιασμού της πρόσβασης της Ευρώπης στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Γι' αυτό το λόγο καλούμε τους εμπειρογνώμονες και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής να συζητήσουν ενεργά τον κανονισμό για τον οπτικοακουστικό τομέα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τη νέα γεωπολιτική κατάσταση. Κατά τη Λετωνική Προεδρία, εμείς θα συμβάλλουμε στη συζήτηση σε σχέση με το μέλλον της οδηγίας ε, περί οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι πρέπει να λειτουργήσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε ε, αυτό που υπάρχει στα συμπερασμάτα της Λιθουανικής και της Ιταλικής Προεδρίας ε, Τέλος, η ενιαία ψηφιακή αγορά δεν μπορεί να αποτελεί μόνο έργο υποδομής και οικονομικό. Κατά κύριο λόγο πρέπει να εστιάζεται στο περιεχόμενο, τη δημιουργικότητα και την ε, πολυμορφία. Ελπίζω λοιπόν να συνεργαστείτε μαζί μου για να μεταφέρουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το μήνυμα. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ήθελα να τονίσω και πάλι θα χτίσουμε μαζί το ευρωπαϊκό μέλλον. Το λογότυπο της Λετωνικής ε, Προεδρίας αποτελεί μάλιστα, είναι μάλιστα η Μιλόπετρα, ε, ένα σύμβολο εργασίας ε, δείχνει την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στον τομέα του πολιτισμού όπως κάνουμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Το σύμβολο της Μιλόπετρας ε, αντικατοπτρίζει τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσετε και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, για τις διαβεβαιώσεις σας ε, για τα θέματα αυτά, τα κεντρικά θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που το ζήτησαν. Θα ξεκινήσω με την Σαμπίν Ράιαν. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, τρία θέματα στα οποία θα ήθελα να εμπαθύνουμε. Πρώτον, πολιτισμός ως τμήμα του κλάδου της δημιουργικότητας. Στο παρελθόν, στα πλαίσια των αναπτυξιακών διαρθρώσεων, συχνά ο τομέας του πολιτισμού, ιδίως στην περιφέρεια, έμεινε απ' έξω. Στην χρηματοδότηση, είτε είναι προγράμματα καθαρά πολιτιστικά που χρηματοδοτούνται, είτε είναι μονάχα είτε είναι πιο έντονος ο οικονομικός χαρακτήρας, τελικά υπάρχουν έργα, σχέδια, τα οποία δεν εντάσσονται σε καμιά από τις κατηγορίες, κατηγορίε, δεν χρηματοδοτούνται ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ούτε από τα πολιτιστικά κονδύλια, ούτε από τα ε, κονδύλια τα καθαρά οικονομικά χρηματοδοτικά, δηλαδή τη βιομηχανία. Γι' αυτό. Το άλλο θέμα είναι το δικαίωμα του δημιουργού και η ψηφιακή οικονομία πάλι υπάρχει εδώ μια παράλληλη κίνηση. Δηλαδή αφενός υπάρχει η αξίωση των καταναλωτών να μπορούν να συμμετάσχουν στην πολιτιστική ποικιλία της Ευρώπης, από την άλλη μεριά η δημιουργία, οι δημιουργοί δηλαδή πολιτισμού θέλουν να μπορούν να επιζήσουν από το επάγγελμά τους. Ερώτημα. Πρόκειται να καταθέσετε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τρίτο θέμα, η συμφωνία με τους Αμερικανούς, τύπ. Υπάρχει εξαίρεση του πολιτισμού μέσα στην διαπραγματευτική εντολή, ωστόσο ξεκάθαρη οριοθέτηση για τα οπτικοακουστικά οδηγεί σε προβλήματα. Ποια εντάσσονται δηλαδή πάλι στην καθαρά οικονομική πλευρά και ποια είναι καθαρά πολιτισμός. Ποια θα είναι η συμβολή εδώ της Λετωνικής Προεδρίας στις διαπραγματεύσεις δηλαδή για την συμφωνία TTIP. Σας ευχαριστώ Σαμπίν. Η Πέτρα Κάμερεβερτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Υπουργέ για τις δηλώσεις σας και για το γεγονός ότι καταστήσατε σαφές ότι η Λετωνική Προεδρία γνωρίζει προπάντων ότι σημαντικό στην Ευρώπη είναι να διατηρηθεί η πολιτιστική ποικιλία, η πολυφωνία των μέσων και των πολιτιστικών συγγνώμη, δημιουργών. Εξ όσων γνωρίζω, η Λετωνική Προεδρία προτίθεται να κάνει προσπάθεια να επιτύχει βήμα προόδου και στην στάση του Συμβουλίου στην ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία πάλι χωρίζεται σε τρία μέρη. Ένα σημαντικό μέρος, το οποίο μας απασχόλησε και στην προηγούμενη θητεία, εδώ εμάς στην Επιτροπή Πολιτισμού δηλαδή, και όπου προσπαθήσαμε να διατυπώσουμε θέσεις του Κοινοβουλίου που τελικώς ευρήκαν και πλειοψηφία, είναι το μέγα θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου. Ουδετερότητα του διαδικτύου είναι μέγιστη τεχνική προτεραιότητα έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η πολυφωνία των μέσων, η πολυφωνία των απόψεων, η δημιουργικότητα, ώστε να μπορέσουν τα έργα πολιτισμού να φτάσουν μέχρι τους τελικούς καταναλωτές. Από όσα ακούω όμως, φαίνεται πως η Λετωνική Προεδρία προτίθεται να κάνει πρόταση όπου η ουδετερότητα του διαδικτύου θα περιλαμβάνεται και θα ρυθμίζεται στον κανονισμό μόνο καταρχήν. Δεν θα της αποδίδεται όμως η σημασία που της έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζήτησε πρώτον να θεμελιωθεί νομοθετικά, δεύτερο να προβλεφθούν και συγκεκριμένοι νομοθετικοί περιορισμοί, υπό οποίου όρους δηλαδή θα μπορούν να είναι δυνατόν να παρέχονται ειδικέ υπηρεσίες. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω εδώ την απόψή σας και πώς εντάσσεστε μέσα σε αυτήν την συναυλία των διαφόρων φωνών υπουργών που αναμειγνύονται όσων είναι δηλαδή αρμόδιοι για πολιτιστικά θέματα. Για τη συμφωνία TTIP θα συμφωνήσω με την προηγούμενη συνάδελφο. Είχαμε ξεκάθαρη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό των οπτικοακουστικών από την εντολή της διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχουν όμως ξεκαθαροί ορισμοί για τον τομέα των οπτικοακουστικών και πρέπει να είναι σαφές ότι η εξαίρεση για τα οπτικοακουστικά μέσα θέλουμε να είναι ευρεία και να είναι γερά θεμελιωμένη για το μέλλον. Να μην περιοριστεί μοναχά στην παροχή υπηρεσιών, αλλά να περιλάβει και τις επενδύσεις στον οπτικοακουστικό τομέα. Γιατί εκεί ενδέχεται να υπάρξει ανοιχτό ένα παράθυρο που να οδηγήσει σε βλάβη και του ίδιου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Διεξήχθη εδώ στην Επιτροπή μας πρόσφατα συζήτηση στα πλαίσια Κροάσεως όπου αναπτύχθηκε η ιδέα ή πάντως συζητήθηκε να ξεκινήσουμε ένα ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς Όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλά έτη με διάφορες ονομασίες. Όπως γνωρίζετε, το, ε, μάλλον αυτό που θέλω να γνωρίζω εγώ είναι αν θα μπορούσατε να υποστηρίξετε την ιδέα αυτή του έτους πολιτιστικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ. Αντινόλφη. Να ευχαριστήσω την Υπουργό. Θα ήθελα να θέσω τρία θέματα Πάνω σε αυτά τα τρία θέματα έχω κάποια ενδιαφέροντα θα έλεγα. Το θέμα της εκπαίδευσης. Όταν συζητάμε τα της εκπαίδευσης δεν την εννοούμε σαν μέσο διανοητικής και προσωπικής κατάρτισης τόσο. Δίδουμε στο σχολείο την υποχρέωση θα έλεγα να αναπτύξει από μόνο του την αίσθηση της ιδιότητας του πολίτη των ε, νέων πολιτών και να οδηγήσει τους πολίτες αυτούς να συλλάβουν και την ίδια την έννοια του έθνους. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, σταθούμε κάπως ε, περισσότερο στα θέματα αυτά ιδιαίτερα στη σχέση που έχουν με την απασχόληση. Νομίζω ότι τα τελευταία γεγονότα, κυρίως αυτά που χτύπησαν την Γαλλία, δείχνουν ότι η άγνοια και η έλλειψη ανοχής οδηγούν αναπόφευκτα στην βία. Η γνώση λοιπόν είναι η βάση της ε, ειρηνικής συμβίωσης και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω τι σχέδια έχετε σαν Προεδρία ε, για να παρέμβετε προς την κατεύθυνση αυτή στον τομέα της εκπαίδευσης. Να ζητήσω επίσης από την Υπουργό να μας πει τι σκοπεύει να κάνει σχετικά με, την, με το μέσο αυτό των εγγυήσεων για τους νέους. Είχε παρουσιαστεί πριν μερικούς μήνες σαν ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο, σχεδόν η πανάκια για όλα τα κακά που χτυπούν τους νέους. Μετά έπεσε σε αφάνεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο φύγει κυρίως τις χώρες του Νότου και ξέρετε ότι οι στατιστικές όχι μόνο δεν δείχνουν βελτιώσεις στις χώρες αυτές, αλλά το αντίθετο. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την Προεδρία αν έχει την πρόθεση να κάνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή και αν έχει κάποια συγκεκριμένα προγράμματα στο νου και τρίτον και τέλος θα ήθελα να σταθώ στον πολιτισμό. Όπως έλεγε και η υπουργό, ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται σαν μια οικονομική κυρίως δυνατότητα και σαν μέσο αύξησης της οικονομικής ευμάρειας. Νομίζω ότι η οικονομική καταρχάς ανάπτυξη δεν συνδέεται υποχρεωτικά με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό έχει διαψευθεί Κάποιες χώρες όπως η Ιταλία και ιδιαίτερα στο νότο της Ιταλίας θα πρέπει να αντιμετωπίζουν και τον πολιτισμό σαν μέσο βοήθειας για την οικονομία και για την απασχόληση. Αλλά δεν θα πρέπει ο πολιτισμός να θεωρηθεί σαν ένα προσπόληση προϊόν. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν ανήκει μόνο σε εμάς αλλά και στις μελλοντικέ γενιές και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει αντικείμενο αξιολόγησης και προστασίας. Σκοπεύετε λοιπόν να αναλάβετε δράσεις έτσι ώστε στο εξάμεινό σας να τονιστεί η οικονομική αυτή σημασία του πολιτισμού. Θα ήθελα να πω ότι θα ακούσουμε την επόμενη ερώτηση και μετά θα πάρουμε μια απάντηση από την Υπουργό και θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ξέρετε ότι αμέσως μετά θα έχουμε και την ακρόαση της Υπουργού Παιδείας, οπότε θα πρέπει να είναι κάπως πιο σύντομη. Τρούπελ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ομιλία σας. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι υποστηρίζω τα όσα υποθήκαν για την ουδετερότητα των δικτύων και για τα όσα είπε η Πέτρα Καμπρεβέρτ για το TTIP. Χρειαζόμαστε ένα σαφή ορισμό για το τι σημαίνει εξαίρεση του πολιτισμού και σαφή ορισμό των υπηρεσιών, των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και επαρκείς αποδείξεις. Έχω τώρα μια ερώτηση προς σας, διότι είπατε ότι η Κομισιόν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, ώστε να διευκολύνονται οι καταναλωτές να έχουν καλύτερη διασυνοριακή πρόσβαση. Αυτό είναι σαφές. Αφενός όλοι έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον, αλλά να σας θυμίσω επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο την αηφόρο χρηματοδότηση του κινηματογράφου. Και το πώ θα βρούμε τη σωστή ισορροπία είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί εδώ. Αλλά θα ήθελα να μάθω και τη δική σα προσέγγιση. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Ακούγονται φήμε ότι πιθανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκέφτεται να εγκαταλείψει την ε, οικονομική υποστήριξη των Ευρωπαίων ε, όπως έχει αυτή τη στιγμή. Θα θέλαμε να μάθουμε την άποψη γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Υπουργό για ένα πρώτο γύρο απαντήσεων ώστε να αποφύγουμε ε, να έχει η υπουργό να απαντήσει σε υπερβολικά πολλές ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. Um, es äh, mēģināšu secīgi Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω με την ίδια σειρά. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσει έγιναν πολύ γρήγορα. Αν ξεχάσω να απαντήσω κάποια από αυτές, θα είναι επειδή δεν πρόλαβα να τη γράψω. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση που αφορά τον πολιτισμό ως δημιουργικό κλάδο και το ότι πολύ συχνά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο πολιτισμός διαχωρίζεται και θεωρείται ότι είναι ξεχωριστός κλάδος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση. Δεν μπορούμε να απομονώνουμε τον πολιτισμό από τους υπόλοιπους κλάδους της ζωής. Γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο μας στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ώστε να αποδείξουμε τη σπουδαιότητα του τομέα αυτού. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτό τον ε, όρο κλειδί, το crossover, τη διασταύρωση αυτή είναι η σωστή προσέγγιση για να δείξουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα και σε άλλους τομείς. Διότι κατά την αποψή μας η συνεργασία είναι ο παράγοντα που θα δημιουργήσει τη δύναμη που χρειαζόμαστε. Δεν πρόκειται να κάνουμε τώρα του κινηματογραφιστές οικονομολόγους ώστε να αξιοποιούν καλύτερα τις οικονομικές διαδικασίες. Είναι σημαντικό απλά για μας αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά του, αλλά και σε συνεργασία με άλλου τομεί γιατί δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος ε, να αναπτύξουν ε, τη δημιουργικότητά τους, τις ιδέες τους, ε, να αποκτήσει νέα αξία ο τομέας τους. Έχουμε πολλά θετικά παραδείγματα ήδη κινήτρων που έχουν δοθεί για καινοτομίε και νέε λύσει. Με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Όχι μόνο στον τομέα τη οικονομία, γιατί πολύ συχνά εστιαζόμαστε μόνο στα οικονομικά. Δεν συζητάμε για την επιπτώση του πολιτισμού στην οικονομία. Πρέπει να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την έννοια του crossover, της διασταύρωσης και ε, με κάποια παραδείγματα θετικά θα μπορέσουμε να δείξουμε ότι οι τέχνες και ο πολιτισμός μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις μεταφορές, την επίλυση των ζητημάτων περιβαλλοντικής αηφορίας, ε, Γι' αυτό τον λόγο κεντρική δραστηριότητα θα είναι η διάσκεψη των εμπειρογνωμόνων με πρωταρχική εστίαση σε αυτά τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό το οποίο και από τις συζητήσεις των προηγούμενων συμβουλίων και που θα συνεχιστεί από τη δική μας Προεδρία και στην επόμενη διάσκεψη του Συμβουλίου το Μάιο είναι το ζήτημα των αποδεικτικών στοιχείων αυτής της επιρροής ε, στην οποία αναφερθήκαμε κατά τη Λετωνική Προεδρία θα συζητήσουμε ε, την έρευνα και την εξέβρεση αποδεικτικών στοιχείων ώστε να δώσουμε ρεαλιστικά αποδεικτικά στοιχεία για το πώς οι τέχνες και η δημιουργικότητα επηρεάζουν θετικά άλλους τομείς. Είχαμε τώρα μια ερώτηση για τη Διατλαντική Συμφωνία εδώ πρέπει, το TTIP, εδώ πρέπει να πω καθαρά τη δική μας άποψη. Μετά από δύο υπουργικά συμβούλια τον Ιούνιο του 2013 και τον Οκτώβριο πέρυσι, μετά από αυτές τις δύο συναντήσεις του Συμβουλίου, θέλουμε να εκφράσουμε μια κοινή άποψη των Υπουργών όλων ότι η οπτικοακουστική πτυχή εξαιρείται από τη Συμφωνία και η Ελληνική Προεδρία υποστηρίζει αυτή την προσέγγιση. Θα υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να, ενημερώσει το Συμβούλιο, να ενημερώνει το Συμβούλιο για το πώς εξελίσσονται οι συζητήσεις αυτές στο μέλλον. Επίσης, ε, ακούστηκε μια ερώτηση από πολλούς, πολλά μέλη, που αφορούσε τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright. Ναι, πράγματι, το ζήτημα του copyright συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Αποτελεί προϋπόθεση για την προσπελασιμότητα, αλλά δεν είναι η μόνη. Διότι όταν μιλάμε για προσπελασιμότητα σε ποικιλόμορφο περιεχόμενο, ε, μεγάλη σημασία αποκτά η τεχνολογική διαλειτουργικότητα. Πολλοί το ανέφεραν. Και επίση και οι διάφορε γλώσσε. Η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι επιλογές, δυνατότητες επιλογής μιας ε, γλώσσας, ενδεχομένω η χρήση της αυτόματης μετάφρασης. Στην ε, διάσκεψη περί οπτικοακουστικών θεματών που θα λάβει χώρα στη Ρήγα το Μάιο, οι εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν αυτά τα ζητήματα και τις ερωτήσεις που κάνατε, θα συζητήσουν και την ουδετερότητα των δικτύων. Σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Συμφωνώ μαζί σας. Η ενιαία ψηφιακή αγορά πράγματι αποτελείται από τρία κομμάτια, τα οποία σχετίζονται στενά και με άλλους τομείς. Γι' αυτό το λόγο έχουμε έναν ειδικό Αντιπρόεδρο πρόεδρο της Επιτροπής ε, που είναι αρμοδίος για αυτούς τους τρεις θεματικούς τομείς. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο, με τον κύριο Επίτροπο Αντιπρόεδρο, ε, θα επιτύχουμε κάποια εναρμονισμένη ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Επίσης, ε, είχαμε μια ερώτηση που αφορούσε το έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική. Προγραμματίζουμε μια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων εστιασμένη στην πολιτιστική κληρονομιά και το πώς αυτή συνδέεται με τη σύγχρονη εκτεκτονική, το design και κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αυτής πιστεύω θα μπορούσαμε να εστιαστούμε σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ για τις πρώτες αυτές απαντήσεις. Παρακαλώ οι δεύτερες ερωτήσεις, η δεύτερη σειρά να είναι πολύ πιο σύντομες. Word, ουδένκα και μετά απαντήσεις. Σύντομα. Yes, I will be very brief. I just wanted to say... Θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, με αυτό το οποίο ακούστηκε ότι ο πολιτισμός είναι η συνείδηση του έθνους. Τώρα έχουμε μια τεράστια μάχη μπροστά μας έτσι ώστε να διατηρήσουμε την ειρήνη και στις χώρες μας και ανάμεσα στις χώρες μας και δεν θα πρέπει ο πολιτισμός να πέσει στα χέρια των ακραίων Αυτός ο τομέας λοιπόν είναι ένας κρίσιμος τομέας, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Και ναι μεν πρέπει να προωθούμε τις, ε, τα πολιτιστικά μνημεία και στοιχεία της χώρας μας, αλλά ταυτόχρονα να μην προωθούμε τη διέρεση και την έλλειψη ανοχής. Βέντα, συγγνώμη. Ευχαριστώ Υπουργέ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Αναφερθήκατε ε, στα θέματα της Προεδρίας σας στον τομέα του πολιτισμού και αναφερθήκατε στο λεγόμενο crossover ε, με θέματα όπως τα ψηφιακά μέσα, η κοινωνική ένταξη κτλ. Η αρχή αυτή του crossover αφορά επίσης και την προώθηση και την υποστήριξη της δημιουργικότητας. Συνεπώς λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας για να προωθήσετε ακριβώς την ευρωπαϊκή αυτή διάσταση σε όλες τις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ συνάδελφε Βέντα. Τελειώσαμε με τον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Υπουργέ πρέπει να απαντήσετε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ιδιαίτερα <clears throat> ε, ενδιαφέροντα μου φάνηκε αυτή για τον κινηματογράφο. Τον Δεκέμβρη στη Λετωνία υποδεχτήκαμε την ε, εκδήλωση απονομής κινηματογραφικών βραβείων πολύ θετικό σημάδι για την διαφήμιση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και στη δική μας χώρα και στην Ευρώπη συνολικότερα και συμφωνώ μαζί σας ότι κάθε προεδρία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, να προβληματιστεί δηλαδή για το πώς θα προωθήσει την κινηματογραφική μας βιομηχανία και τις κινηματογραφικές ταινίες ως έργα τέχνης. Η Ευρώπη είναι ενωμένη στην πολυμορφία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Προεδρία έχει την ευθύνη μέσω των δραστηριοτήτων της να τονίζει την ποικιλομορφία, την πολυφωνία των ευρωπαϊκών έργων τέχνης. Βέβαια θα μιλήσουμε και για κινηματογράφο στην ε, διάσκεψη που θα οργανώσουμε για την διασταύρωση μεταξύ των πολιτιστικών ρευμάτων, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο κινηματογράφος και για, την, και για θέματα παιδείας, αλλά και για να ρίξει φως σε ορισμένες κοινωνικές καταστάσεις. Έτσι ανδρώνεται ο πολιτισμός και μέσα από τα οπτικοακουστικά μέσα σημαίνει ότι μπορούμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για ένα επίκαιρο θέμα στην κοινωνία και ο κινηματογράφος είναι καλό παράδειγμα αυτού του crossover με την έννοια στην οποία αποδώσατε και εσείς. Στις προηγούμενες απαντήσεις μου, στις ερωτήσεις μου, δεν, ε, μίλησα στην κυρία, δεν απάντησα στην κυρία Αντινόλφη για τις συνέργειες. Συμφωνώ ότι ένας τύπος συνέργειας μεταξύ πολιτισμού και παιδείας είναι αυτός που δίνει περιεχόμενο στην παιδεία. Και άλλωστε η παιδεία είναι ο καλύτερος τρόπος για να διδάξει κανείς τις αξίες. Και από την άλλη μεριά η παιδεία προσφέρει και το μέσον για την πρόθεση των πολιτιστικών αξιών. Είμαι βεβαία ότι και η συνάδελφός μου, η Υπουργός Παιδείας, θα τα εξηγήσει ακόμα καλύτερα. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σα ότι χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη συνέργεια, συνεργασία δηλαδή μεταξύ παιδεία και πολιτισμού. Πρέπει να μιλήσουμε για πολιτισμό, πρέπει να μιλήσουμε για αξίες, πρέπει να μιλήσουμε για ανοχή. Τι σημαίνει ανοχή, πώ εννοείται η ανοχή. Αυτά θα τα βάλουμε και πίσω ως θέματα και στην διάσκεψή μας. Και θα δώσουμε και ορισμένα θετικά παραδείγματα από την ίδια τη Λετωνία, όπου έχουμε τώρα πιλωτικό πρόγραμμα για τη συνεργασία μεταξύ παιδείας και πολιτισμού. Και αυτά θα τα περιλάβουμε, όπως είπα, και σε μια από τις διασκέψεις που θα, οργανώσουμε. Erasmus on Europeana uh, uh, Είχατε καμιά ερώτηση για το πρόγραμμα Ευρωπαϊάνα. Τα νεσαντζερδέα, βα ιούς βαράτε λούτζα ατκάρτουτ. Κας τιμς τίεσαι ίντρεσε Ευρωπαϊάνα κόντεκ. Δεν άκουσα την ερώτηση. Δεν άκουσα την ερώτηση. Τι ακριβώς είπατε για αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχουν φήμες ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η χρηματοδότηση του Ευρωπαίαν ή τέλος πάντων υπό τη μορφή την οποία έχει αυτή τη στιγμή. Έχετε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό, αναλαμβάνετε κάποια δέσμευση. Ε, ποια είναι η τελο παντων υπο τη μορφη την οποια εχει αυτη τη στιγμη εχετε κάποια πληροφοριες γι αυτο αναλαμβανετε καποια δεσμευση ποια ειναι η προσεγγιση σας για το θέμα αυτό. Jā, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. paldies, es tagad sapratu jūsu jautājumu, ναι, τώρα κατάλαβα την ερώτησή σας. Απογοητεύομαι που ακούω κάτι τέτοιο, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τέτοιες φήμες. Είναι απαράδεκτο. Εδώ στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργαστούμε για να συνεχίσουμε αυτό το εξαιρετικό έργο. Βάσει των πληροφοριών που έλαβα εγώ το 2014, το Ευρωπαϊκό παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 33 εκατομμύρια πολιτιστικά αντικείμενα σε 500 σημεία στην Ευρώπη. Και αυτή η πρόσβαση σε ένα τόσο ευρύ ε, πόρο πολιτισμού και παιδείας είναι κάτι μοναδικό. Όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να υποφεληθούν αυτό. από αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παιδεία όλων των ηλικιών. Ως Προεδρία εμείς ε, θα συνεργαστούμε μαζί σας σε οποιασδήποτε συζητήσεις που θα αφορούν τη διατήρηση της χρηματοδότησης του προγράμματος αυτού. Um, Ευχαριστώ την Υπουργό. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, αν θέλει να κάνει κάποιες ε, διευκρινήσεις. Θυμίζω ότι αύριο έτσι και αλλιώς θα έχουμε και την ε, συνάντηση με τον Επίτροπο. Μπορείτε να μας δώσετε μια κάποια πρώτη απάντηση στην παρούσα φάση. Σύντομα παρακαλώ, Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, parole pour discuter les priorités. No. In questo caso no, è una richiesta che viene dalla Commissione, non dalla Presidente. Λοιπόν, είναι η ερώτηση που τέθηκε από την Επιτροπή μας, όχι από την Προεδρία. Μπορείτε να κάνετε μια διευκρίνηση, θα έλεγα. Επιμένω. Yes, thank you, madam. Madam. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τη Λετωνική Προεδρία που εξήγησε ποιος είναι ο σχεδιασμός της για τους επόμενους έξι μήνες. Βεβαίως εμείς υποστηρίζουμε και όλες τις ιδέες που ανέφερε και με την ευκαιρία θα ήθελα επίσης να ανακοινώσω ότι ο, αύριο θα είναι παρόν ο, Υπουργό, ο, Επίτροπος στην παρούσα Επιτροπή και νομίζω ότι το καλύτερο θα είναι ο ίδιος ο Επίτροπος να σχολιάσει τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ακούσω, ότι αύριο θα τεθεί το θέμα αυτό από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Επίτροπο μάλλον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, είμαστε ικανοποιημένοι από τη σημασία την οποία δίδεται στα θέματα τα οποία μας αφορούν ιδιαίτερα την αναθεώρηση της στρατηγικής 2020 γύρω από τον πολιτισμό, γύρω από το ραδιοτηλεοπτικό μέσο, γύρω από την ψηφιακή αγορά και βλέπουμε ότι θα γίνει μια προσπάθεια την οποία θα παρακολουθήσουμε και στην οποία θα συνεισφέρουμε. Και γι' αυτό ακριβώς ε, φέραμε την προσοχή σας και εξετάζουμε και εμείς ήδη την δυνατότητα να δημιουργήσουμε γέφυρες ανάμεσα στον προϋπολογισμό και τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές όπως την οικονομία και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες οι οποίες μπορεί να υπάρχουν για την χρήση των πιστώσεων αυτών, των δυνατοτήτων των οικονομικών τις οποίες έχουμε μέσω του Horizon, μέσω κάποιων άλλων επιμέρους προγραμμάτων, έτσι ώστε να φέρουμε πάρα πολύ κοντά την πραγματική οικονομία στον πολιτισμό. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά, λέει η Πρόεδρος, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ενέργειές σας και την πολιτική σας σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσδοση πολιτισμικής διάστασης στην ψηφιακή αγορά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή δουλειά. Eh, Ωραία, συνεχίσουμε με την Υπουργό Παιδείας και Επιστημών, την κυρία Μαρίτε Σέιλε, η οποία θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Ε, είδατε κάπως πώς οργανώνουμε τις εργασίες μας ε, μέχρι στιγμής. Ε, θα κάνουμε το ίδιο όπως και πριν. Θα σας δώσουμε κάποιο χρόνο. Ε, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Siamo molto felici di averla qui. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε εδώ. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία όπως προηγουμένως. Ε, όπως είδατε προηγουμένως, ε, θα... μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσουμε και από εσάς τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας, όπως έχουμε ήδη δει, θεωρούμε πολύ ενδιαφέρουσε. Μας ενδιαφέρει ότι εστιάζεστε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το επόμενο εξάμεινο της Προεδρίας σας, ειδικότερα για την επανεκκίνηση ε, της, για την εκ νέου της ε, ατζέντα για την απασχόληση, ε, για τις εταιρικέ σχέσεις, τα partnership που θέλετε να ενισχύσετε. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικός και ο ρόλος που θα παίξετε και βάσει μιας από τις προτεραιότητες της Κομισιόν για το νέο επενδυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει την παιδεία ως μία από τις πέντε προτεραιότητες. Παρότι στα δέκα σημεία ε, των προτεραιοτήτων του κυρίου Γιούνκερ δεν υπάρχει ιδιαίτερα η λέξη παιδεία. Υπολογίζουμε λοιπόν στη Λετωνία ε, για να εστιαστούμε περισσότερο σε αυτό το θέμα ε, και για να τηρηθούν και οι προθεσμίες που έχουμε μέσα στο επόμενο πεντάμενο. Έχετε τον λόγο, θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή. Αξιότιμη Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή και σημαντικό έργο για μένα το να προσθέσω τις προτεραιότητες της Λετωνικής ε, Προεδρίας. Πιστεύω ότι αυτό θα ενισχύσει τις σχέσεις μας και θα συνεχίσω τώρα στα λετωνικά. mūsu prezidentūras trio partneru Έχουμε σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη την συνεργασία με τους εταίρους μας της Τριάδος των άλλων δύο προεδριών δηλαδή. Έχουν αρχίσει οι εργασίες μας. Με μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Προεδρίας μας για την παιδεία, νεότητα και αθλητισμό. Η Λετωνική Προεδρία θα τονίσει ιδιαίτερα τον όρο της παιδείας για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πρόθεση των επενδύσεων, για την διευκόλυνση της εξέβρεσης απασχόλησης και την ευμερία των ανθρώπων γενικότερα. Με, μέσα στα πλαίσια της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της, το θεματολόγιο της παιδείας και εκπαίδευσης χρειάζεται νέα όθηση είναι δυνατό με στενότερες συνέργειες μεταξύ της Στρατηγικής Ευρώπης 2020 και του Στρατηγικού Πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία, Εκπαίδευση και Παιδεία, να γίνει λοιπόν η συνεργασία αυτή. Η Λετωνική Προεδρία θα προωθήσει συζήτηση για τα κέρια στοιχεία, key elements, του στρατηγικούς στόχους και την διαχείριση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της παιδείας, συμβάλλοντας έτσι στην σύνταξη της κοινή έκθεσης για το 2015. Θα παρακολουθούμε βεβαίως πολύ προσεκτικά τις συζητήσεις που διεξάγονται στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερο, η Λετωνική Προεδρία θα συνεχίσει το έργο της στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Θα λάβουμε υπόψη βεβαίω και, τους, και τις νυν και τις μελλοντικέ προκλήσεις. Θα προωθήσουμε τη συζήτηση για το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης με βασικό στόχο να ενισχύσουμε τη συνεργασία των χωρών μελών, των κοινωνικών εταίρων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε αυτοί να γίνουν ανταγωνιστικοί στις αγορές απασχόλησης και για να μπορέσουν εν τέλει να αναπτυχθούν και προσωπικά. Η Λετωνική Προεδρία σχεδιάζει συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Αρμοδίων για Επαγγελματική Κατάρτιση Κοινωνικών Εταίρων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ρήγα στις 22 Έκτου για να συζητήσουμε για περαιτέρω κοινού στόχους και καθήκοντα στα πλαίσια της σχετικής ανακοίνωσης. Εκτός από αυτό, η Προεδρία θα προωθήσει την παραπέρα διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό θα γίνει με ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών. Θα οργανώσουμε την 5η ΑΣΕΜ στην Ρήγα στις 27 και 28 Τετάρτου. Εκεί θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα που θα έχουν επιτευχθεί από την προηγούμενη ε, Υπουργική προ, προ δύο ετών. Οι Υπουργοί θα καταστρώσουν στόχους για το μέλλον για να σφυριλατηθεί στενότερη περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων στις περιφέρειες. Από τότε που ξεκίνησε το 1999 η διαδικασία της Μπολόνια, οι βασικοί στόχοι δεν έχουν αλλάξει. Η δημιουργία απλού και συγκρίσιμου συστήματος πτυχίων είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να διασφαλίζονται τα αποτελέσματα και η ποιότητα της εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας Αναμένουμε να γίνει αξιολόγηση της διαδικασίας της Μπολόνια φέτος σε συνδυασμό με την διάσκεψη των Υπουργών Αρμόδιων για Μπολόνια που θα γίνει στο Γερεβάν της Αρμενίας για να προχωρήσει η ανάπτυξη, να μειωθεί η ανεργία, να ενισχυθεί η μελλοντική ευημερία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την καινοτόμα της ικανότητα και να προσφέρει ευκαιρίες στους νέους. Γιατί οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν με τρομερή ταχύτητα πλέον τις ζωές μας. Οι πιο επιτυχημένες περιφέρειες θα είναι στο μέλλον εκείνες οι οποίες έχουν κατοίκους που είναι ενήμεροι για την ψηφιακή τεχνολογία και ικανοί να την χειριστούν. Αναγνωρίζουμε ότι η προσχολική εκπαίδευση καθώς επίσης η στοιχειώδεις, είναι ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη των παιδιών. Γι' αυτό η Προεδρία μας σχεδιάζει να συζητήσει τον ρόλο των ε, περιόδων αυτών της σχολικής ζωής για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων. Η Προεδρία, σε συνεργασία με τις χώρες μέλη, αναγνωρίζει ότι χρειάζονται εξειδικευμένες λύσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας της παιδείας, θα αρχίσουμε συζήτηση και για την προσβασιμότητα της παιδείας. Εκτός από αυτό θα προωθήσουμε τη συζήτηση για την διαφάνεια και την αναγνώριση των προσόντων, πτυχίων και προσόντων, και των μελλοντικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, λαμβάνοντα υπόψη ότι οι υπάρχουσες προκλήσεις μειώνουν τη δυνατότητα απασχόλησης και προκαλούν εμπόδια στην κινητικότητα. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε καλύτερη ισορροπία μεταξύ δεξιοτήτων και εργασίας και ενίσχυση επομένως της ανταγωνιστικότητας. Αξιότιμα μέλη, συνεχίζοντας, επιθυμώ να τονίσω ότι οι νέοι άνθρωποι είναι πολύτιμο δυναμικό και μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της Ευρώπης. Ας μην το λησμονούμε αυτό. Αυτή ας είναι η βάση της εργασίας μας. Ας προσφέρουμε στους νέους τη δυνατότητα να αναπτύξουν το δυναμικό τους πλήρως. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορθά τις προκλήσεις πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους να αντιμετωπίσουν και αυτοί με τις σειρά τους τις προκλήσεις, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασής τους ε, που έχουν ληφθεί είναι σημαντικά, εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπίλητα προβλήματα, τα οποία έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση των νέων στην Ευρώπη. Προκαλούνται προβλήματα από την μακρού χρόνο ανεργία και από την έλλειψη ενθουσιασμού που συνεπάγεται αυτή. Οι νέοι συχνά δεν διαθέτουν τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να περάσουν από τη σχολική ζωή στην επαγγελματική. Εάν δεν αντιμετωπιστούν σωστά οι βασικές ανάγκες των νέων, θα οδηγηθούμε σε πολύ βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα. Παρόλο που η μείωση της ανεργίας των νέων είναι πρώτη πολιτική προτεραιότητα στην Ευρώπη, το δυναμικό της ε, πολιτικής αυτής δεν το εκμεταλλευόμαστε επαρκώς. Για να βελτιώσουμε τις μελλοντικέ προοπτικές των νέων, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των τομέων της απασχόλησης, της παιδείας, της κοινωνίας, της κοινωνικής υγείας, δηλαδή της κοινωνικής πρόνοιας και ούτε καθεξής. Αυτά είναι ουσιαστική σημασία για να οδηγηθούμε σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων. Η Λετωνική Προεδρία πιστεύει ότι η νεότητα μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που θα επιτρέψουν με τη σειρά τους, εφόσον επιληθούν, την ανάπτυξη προσωπικότητας των ατόμων και την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες και για την απασχόληση. η ανάπτυξη προσωπικότητας αναπτύσσει και την αρχή, την ανεκτικότητα των ανθρώπων μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό για τους νέους αυτό. Είμαστε πεπισμένες ότι τα θέματα της νεότητας πρέπει να περιληφθούν και σε άλλους τομείς πολιτικής και σε άλλους χώρους της πολιτικής για να μπορέσουν έτσι να επιληθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα η Λετωνική Προεδρία θα ρίξει ιδιαίτερο φως στην διατομιακή συνεργασία για να προσφέρει πιο αποτελεσματικές λύσεις στους νέους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματά τους. Θα προωθήσουμε δε και συμπεράσματα για το Συμβούλιο Υπουργών του Μαΐου, μάλλον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαΐου, για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας και να ενισχύσουμε και την απασχόληση αλλά και την απασχολησιμότητα θα οργανώσουμε το δεύτερο φόρουμ νεολαίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας. Είναι επεπισμένη η Προεδρία μας ότι η συνεργασία με τους νέους είναι ο καλύτερος τρόπος για να τους στείλουμε χείρα βοηθείας. Για να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται κοινωνικά αποκλεισμένοι. Η πολιτική υπέρ των νέων μπορεί να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και λαμβάνοντα υπόψη τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 που έχει μηχανισμούς εφαρμογής αλλά και οδικό χάρτη και μετά από μια ενδιάμεση αξιολόγηση ως κύριο στόχο θα έχει να συμβάλλουν οι νέοι στην εκπλήρωση κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Η Λετωνική Προεδρία τονίζει ότι η πολιτική νεολαίας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση των στόχων της Ευρώπης 2020. Θα περιληφθεί άλλωστε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου. Ο διαρθρωμένος διάλογος είναι σημαντική διαδικασία και ο διαρθρωμένος διάλογος έχει ως στόχο την ενίσχυση των προτεραιοτήτων της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής για τους νέους. Στην διάσκεψη που θα διεξαχθεί στην διάρκεια της εβδομάδας νέων, η νεολαίας, θα έρθουν σε επαφή πολλές χιλιάδες νέων με αυτούς που ασκούν την πολιτική, policy makers δηλαδή, Ήδη η διαδικασία διαβουλεύσεως έχει διαρκέσει ένα πεντάμινο και η διάσκεψη του Μαΐου θα γίνει στη Ρήγα. Μάρτιο καλύτερα. Θα γίνει 24 με 26 Μαρτίου στη Ρήγα με συμμετοχή νέων και ω θέμα θα έχει τη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Ευρωπαρόμετρο μόνο 20,8% των νέων που έχουν δικαίωμα ψήφου συμμετέσχαν στις ευρωεκλογές. Έχει κέρια σημασία να, να σπρώξουμε τους νέους να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή της Ευρώπης. Στο Συμβούλιο του Μαΐου θα καλέσουμε τους υπουργούς να συζητήσουν την εμπλοκή στα πολιτικά των νέων, στην πολιτική ζωή. Συνεχίζει στα αγγλικά να μιλήσω τώρα, α, πάλι λετωνικά, για τον, για αθλητισμό. Ο λαϊκός αθλητισμός είναι ένας δημοφιλής τρόπος απασχολήσεως, αλλά προσφέρει και ιδιαίτερη, ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία, διότι βελτιώνει την υγεία και ούτω καθεξής. Ο λαϊκός αθλητισμός οδηγεί σε μια θετική στάση του κοινού απέναντι στα προβλήματα της ζωής και ενισχύει τις ε, ικανότητες του καθενός. Και διατομιακές ικανότητες μάλιστα, εφόσον ο αθλητισμός είναι οργανωμένος, αλλά και στον απλό αθλητισμό στους δρόμους. Πολύ σημαντικός αθλητισμός, ιδίως για τους νέους, και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα βέβαια της γύρανσης του πληθυσμού να μπορούν ε, να ε, χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες που αποκτούν μέσω του αθλητισμού και σε διάφορους άλλους τομείς. Πρέπει να δούμε πώς μπορούν τα διάφορα αθλήματα να αναπτύξουν και άλλες ικανότητες, κοινωνικές ικανότητες, τρόπους επιλύσεως προβλημάτων, ε, επαφής με άλλους, την ικανότητα να λειτουργεί κανείς ως μέλος μιας ομάδας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τους νέους. Η Λετωνική Προεδρία λοιπόν σχεδιάζει να συντάξει συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση του αθλητισμού για την ανάπτυξη πολυτομιακών ικανοτήτων, ιδίω για του νέου. Επειδή είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό, η Λετωνική Προεδρία θα οργανώσει μάλιστα και διάσκεψη με τίτλο Αθλήματα και αθλητική δραστηριότητα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Πάλι αυτό θα γίνει στη Ρήγα θα συνεχίσει και τις συζητήσεις η Λετωνική Προεδρία για την πρόθεση των αθλητικών δραστηριοτήτων, των σωματικών αθλημάτων και αυτό θα καταλήξει στον Μάιο στο Συμβούλιο Υπουργών που θα προχωρήσει σε συζήτηση πολιτικής όπου οι υπουργοί των χωρών μελών της Ένωσης που είναι αρμόδιοι για τον αθλητισμό να αναπτύξουν απόψεις για τις καλύτερες στρατηγικές για την πρόθεση των ε, αθλητικών ικανοτήτων. Σε πολλά αθλήματα μάλιστα βλέπουμε και πολλά σκάνδαλα τα οποία οδηγούν σε χειραγωγήσεις αγώνων κλπ. Το τελευταίο σκάνδαλο μάλιστα είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, το είδαμε αυτά στον τύπο. Όμως παρόμοιες περιπτώσεις είδαμε και σε πολλά άλλα αθλήματα και σε διάφορες χώρες μέλη. Η Λετωνική Προεδρία θα παρακολουθήσει και τις διεθνείς εξελίξεις για τα στημένα, τους στιμένους αγώνες. Μάλιστα υπάρχει και η σύμβαση για την αντιμετώπιση του λεγόμενου match fixing που είναι ανοιχτή για υπογραφές. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία της Κομισιόν θα προωθήσουμε προτάσεις για την κύρωση της ε, σύμβασης αυτής και μάλιστα αυτό είναι και πολύ υψηλή προτεραιότητα για μας. Σύμφωνα με τις οικίες ε, διατάξεις της συνθήκης, η Προεδρία, το Συμβούλιο, θα διαβουλευτεί και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Επίσης για το σκάνδαλο του ντόπινγκ, για τα σκάνδαλα του ντόπινγκ. Η Λετωνική Προεδρία θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος σε θέματα αντι-ντόπινγκ, γιατί είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιταχθεί στεναρά στο ντόπινγκ με σταθερή συνεργασία και με μια ενιαία έκφραση. Όταν θα συναντώμεθα και μέσα στα πλαίσια, με ενιαία φωνή δηλαδή να μιλούμε, μέσα στα πλαίσια του Διεθνού Οργανισμού που συνεχίζει το έργο του και βεβαίω και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα παρουσιαστεί από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τον Μάιο στην διάσκεψη του οργανισμού Anti-Doping το Μάιο φέτος. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μου και είμαι βεβαίως στην διάθεσή σας για να ακούσω τις ερωτήσεις σας και βεβαίως επίσης είστε καλοδεχόμενοι να συμμετάσχετε και στι διάφορες εκδηλώσεις που θα οργανώσει η Εντετονική Προεδρία. Ευχαριστούμε κυρία Σέιλε για την ομιλία σας. Ευχαριστούμε που μιλήσατε τόσο καθαρά, προσθέστε με τέτοια καθαρότητα αυτές τις προτεραιότητες. Μάλιστα, εμείς έχουμε δεσμευτεί, δεσμευτεί σε μεγάλο βαθμό για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς. Τελείτου του επόμενου μήνα έχουμε μάλιστα μία ακρόαση στην Επιτροπή Απασχόληση για θέματα που αφορούν τη βελτίωση τη παιδεία και τη απασχολησιμότητα των νέων. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση. Να αναφερθώ και στην έκθεση που θα παρουσιάσουμε μετά, όπου έχουμε συνομιλωτή ε, συνομιλητέ και άλλε επιτροπέ που αφορά τη διαδικασία τη Μπολόνια. Μα ενδιαφέρει η ενίσχυση τη διεθνοποίηση. Μα ενδιαφέρει και αυτή η εταιρική σχέση που θέλετε εσεί να προωθήσετε στο πλαίσιο τη ΑΣΕΑΝ με τις χώρες από Και αυτό φυσικά το τελευταίο θέμα του αθλητισμού είναι κάτι που τέθηκε και στην ακρόαση. Ερώτημα που τέθηκε προς τον Επίτροπο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπογράφει ε, την ανακοίνωση για τον αθέμητο ανταγωνισμό, συναγωνισμό, τον ντόπινγκ, όλα αυτά τα στοιχήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε θα αποτέλεσουν αντικείμενο συζήτηση, την οποία εγώ τώρα. Έχουν ζητήσει το λόγο τρει συνάδελφοι. Δεν ξέρω κάποιο άλλο αν θέλει κάτι. Ε, ε, πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε ορισμένα από τα θέματα. Αφενός ανεργία των νέων και εφαρμογή, εκτέλεση δηλαδή, της εγγύησης νέων. Υπάρχουν διάφοροι τομείς όπου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία αφενός η ανώτερη εκπαίδευση αλλά και η πρακτική επαγγελματική κατάρτιση, vocational training. Σε ορισμένες χώρες μελή υπάρχει το σχολικό σύστημα, αλλού υπάρχει ένα διτό σύστημα που προβλέπει και συνεργασία και μεταξύ των ανωτάτων σχολών αλλά και των επαγγελματικών σχολών και της βιομηχανίας και αυτό τονίζεται ιδιαίτερα ως θετικό χαρακτηριστικό για να επιτρέψει και την μετάβαση από την σχολική ζωή στην επαγγελματική. Έχει αποδείξει την αξία του αυτό το σύστημα. Βλέπετε τη δυνατότητα να προωθηθεί και για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις το σύστημα αυτό μέσα στα πλαίσια της Λετωνικής Προεδρίας. Να υποστηρίξετε δηλαδή το θέμα, το, να υποστηρίξετε την προσέγγιση αυτή, αυτό το dual system και μέσα στα πλαίσια της εγγύησης της νεολαίας. Άλλο θέμα διαδικασία της Μπολόνια. Είπατε ότι στην διάσκεψη της Ρήγας θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής. Θα γίνει και μια αξιολόγηση για το πώς έχει προχωρήσει δηλαδή η διαδικασία της Μπολόνια. Για μένα μπαίνει το θέμα πάντα ότι τα διάφορα ανώτατα ιδρύματα αναγνωρίζουν καμιά φορά τα credit points των διαφόρων κύκλων σπουδών, άλλες φορές όμως όχι. Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο θεωρητικό μοντέλο bachelor και master και από τη μια μεριά και στην πρακτική του εφαρμογή από την άλλη. Κάτι το οποίο οδηγεί σε σημαντικές δυσκολίες στην κινητικότητα των σπουδαστών. Το ίδιο και για τα τελικά πτυχία των σχολών που εξακολουθεί σε πολλές, σε πολλές χώρες να είναι προβληματικό. Ακόμα δηλαδή και όταν λάβουν το, πτυχία, το πτυχίο τους από ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε μια χώρα μέλος δεν αναγνωρίζεται αλλού. Και ιδίω όταν πρόκειται για διδακτορικά και άλλα σχετικά. Ένα άλλο θέμα όπου θέλω να ακούσω κάπως περισσότερα από εσά είναι το ζήτημα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός προβλέπεται εκεί είναι πάρα πολύ μικρός. Πιο συγκεκριμένα, τι βήματα θα κάνετε μέσα στα ε, πλαίσια της, της Λετωνικής Προεδρίας. Έτσι ώστε να προωθηθεί η μη τυπική εκπαίδευση, αλλά και να αναγνωριστεί ιδίως. Σας ευχαριστώ. Τσβέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή την οποία μας παρουσιάσατε. Νομίζω ότι ασχοληθήκατε με τα πιο σημαντικά από τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε κάποια από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε η συνάδελφος πριν από μένα. Στην Ευρώπη έχουμε ένα θέμα σχετικά με τα συστήματα εκπαίδευσης. Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε τα θέματα του πολιτισμού μακράν των οικονομικών παραγόντων και μακράν της παραγωγικής διαδικασίας. Κάποιες χώρες είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά πολλές δεν είναι. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να φέρουμε κοντά τα συστήματα της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες, αλλά θα ήθελα και τις δικές σας απόψεις. Μπορούμε άραγε να συμπεριλάβουμε περισσότερα στοιχεία από την αγορά εργασίας στο πεδίο της, της εκπαίδευσης. Σε κάποιες χώρες επαναλαμβάνω αυτό γίνεται, αλλά θα πρέπει να γίνεται και σε περισσότερες. Και ποια είναι η άποψή σας για την μεταρρύθμιση της διαδικασίας Μπολόνια. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι το παλαιότερο σύστημα είναι καλύτερο και αυτό το πιστεύουν και πολλοί φοιτητέ, αλλά κυρίως και πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί. Εάν η Ευρώπη θέλει να είναι περισσότερο ανταγωνιστική θα πρέπει να αποδειχθεί θα έλεγα την φιλοσοφία των πανεπιστημίων της ε, τρίτης γενεάς. Πανεπιστημίων όπως το Βεσάλιους που είναι πανεπιστήμια καινοτόμα και τα οποία δεν εξαρτώνται κυρίως από την χρηματοδότηση των κυβερνήσεων και του δημοσίου. Λοιπόν, άκουσα ότι θέλετε να ενδιαφερθείτε ε, για τα σωστά θέματα. Άκουσα σε αυτά που είπατε και διέκρινα έναν κάποιο ενθουσιασμό και αυτό μου άρεσε. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι για τους επόμενους πέντε μήνες μαζί θα κάνουμε σημαντικά βήματα. Ευχαριστώ κύριε Τσβέρ. Διακόνου. Merci. Ε, Ευχαριστώ, Υπουργέ. Αυτά τα οποία είπατε ε, νομίζω ότι είναι χρήσιμα και επί της ουσίας και επί της μορφής. Τι εννοώ με αυτό. Δίνεται την δυνατότητα να ξεκινήσει για μια ακόμη φορά μια συζήτηση. Για μια ακόμη φορά όμως. Νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προεδρίας της Ιταλικής το ίδιο είχαμε πει. Ο υπουργό Πολιτισμού είχαμε ακριβώς, είχε ακριβώς τις ίδιες θέσεις και επιθυμίες με τις δικές μας. Και εδώ είναι το θέμα του να εξηγήσει κανείς την διαφορά ευτυχίας και δυστυχίας σε ένα νέο ο οποίος τώρα ξεκινά την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Νομίζω ότι η έλλειψη επιθυμίας ακριβώς των νέων στη συγκεκριμένη εποχή οφείλεται στην έλλειψη δυνατοτήτων για το τι μπορεί να πετύχουν. Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός νέου ο οποίος ξεκινά την επαγγελματική του ζωή. Πηγαίνει σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια σχολή εξειδικευμένη, ε, πολλά του υπόσχονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, φτάνει στο τέλος και εκεί χτυπάει σε ένα τείχο. Εκεί η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη και υψηλότερη από ό,τι περίμενε. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στη δική μου χώρα δυστυχώς. Ε, πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα πανεπιστήμια σαν παράδειγμα που τίνει στην απόκτηση περισσότερων φοιτητών έχει κάποιο νόημα. Φοβάμαι ότι παρουσιάζει κινδύνους μια τέτοια αντίληψη γιατί τελικά πολλοί από τους νέους που ε, έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα πολλές φορές είναι όχι απλά διπλωματούχοι αλλά πολλοί διπλωματούχοι των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και αυτό δεν τους βοηθά σε τίποτα. Συνεπώς λοιπόν αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να δούμε ε, τι θα γίνει για το θέμα του ανταγωνισμού των πανεπιστημίων. Έχει γίνει άλλωστε και μία μελέτη και περίμενα να μεταφραστεί και στην δική μου γλώσσα για να την παρουσιάσω ε, στα πανεπιστήμια μου και στην κυβέρνησή μου, στον Υπουργό Παιδείας. Το θέμα δεν είναι να μην δείξουμε ένα-δύο σωστές πρακτικές από κάθε εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το θέμα είναι να τα συνδυάσουμε και να τα συγκεντρώσουμε για να αποκτήσουμε μια σωστή εικόνα των ορθών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μόνο θα μας επιτρέψει νομίζω να καταλήξουμε σε ε, θετικά στοιχεία για τους ε, Ευρωπαίους φοιτητές και έτσι θα μπορέσουμε να καταστήσουμε και κάθε επαγγελματική δραστηριότητα αξιοπρεπή, γιατί μην ξεχνάτε κάποιες απαράδεκτες νοοτροπίες οι οποίες λέγουν ότι ένα επάγγελμα είναι αξιοπρεπές και ένα άλλο όχι. Ποιος μπορεί να κάνει την αλλαγή εδώ, το σχολείο, το πανεπιστήμιο. Ελπίζω σε έξι μήνες να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ευχαριστώ συνάδελφε Διακόνου. Η συνάδελφος Αντινόλφη. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ να κάνω την ίδια ερώτηση προς την κυρία Υπουργό για την εγγύηση για τους νέους. Το έργο αυτό φορά το πρόβλημα της ανεργίας. Ε, πώς ξαφνικά λοιπόν εξαφανίστηκε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, έχουν διαπιστωθεί, έχουν δημοσιευτεί, έχουμε κάποια νέα από αυτό το πρόγραμμα, κατά πόσο πέτυχε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Επίσης, ε, εσείς ως Προεδρία θα συνεχίσετε στην ίδια οδό ή θα προτείνετε κάτι νέο. Και μετά κάποια μικρή σκέψη. Κατά την άποψή μου, η ενεργεία των νέων δεν οφείλεται πάντα στην επαγγελματική κατάρτιση. Γιατί έχει παρατηρηθεί, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις ε, παιδιών που έχουν κατάρτιση, όχι απαραίτητα ε, προσανατολισμένοι σε τεχνικές εργασίες και παρόλα αυτά ε, στη Βόρεια Ευρώπη και παρόλα αυτά απορροφώνται από τις αγορές της Βορειάς Ευρώπης. Έβλεπα τα στοιχεία του 2013 όσον αφορά τη χώρα μου. Έχουμε τεράστια ροή ατόμων από τον νότο προς το βορρά της Ευρώπης. Να ρωτιόμουν λοιπόν και ρωτώ και την κυρία Υπουργό Κατά την άποψή σας, αυτή η σταθερή ροή νέων μεταναστών αν επεκταθεί στο μέλλον θα δημιουργήσει ανισορροπίες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνάδελφος κύριος Βέντα. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για τα λόγια σας για τον αθλητισμό. Με ενδιαφέρει πολύ αυτός ο τομέας, ε, από αυτόν προερχόμαι. Ναι, συμφωνώ. Όλοι γινόμαστε υγιέστεροι αν κάνουμε... Ε, θα και ευχαριστούμε που αναφέρατε και τα ζητήματα των στημένων παιχνιδιών, όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στον αθλητισμό. Υπάρχουν δύο τύποι αθλητισμού, ο αεραστεχνικός και ο επαγγελματικός. Ε, οι αεραστέχνες φυσικά θα ήθελαν να γίνουν επαγγελματίες και να γίνουν αθλητικοί ήρωες, αλλά δυστυχώς ε, αυτό δεν ε, είναι δυνατόν επιτευχθεί από όλους. Αυτή η διπλή φύση της αθλητικής παιδείας και της απόκτησης δεξιοτήτων θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Προεδρία σας. Ε, θα αποτελέσει και κομμάτι της ε, εκπόνησης ε, επαγγελματικού, επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων πώς θα γίνει να αποφύγουν αυτοί οι άνθρωποι αυτούς τους κινδύνους όπως τα στημένα παιχνίδια. Πώς θα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ε, ο κάθε επίδοξος αθλητής ακολουθεί τη σωστή οδό για τη σωστή εκπαίδευση. Ε, ευχαριστούμε. Παρακαλώ κύριο Σέκοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Σέλ, κατανοήσατε ποια είναι τα προβλήματα που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι όμως να μείνουμε στην αναγνώριση των συμπτωμάτων, αλλά στην θεραπεία τους. Ε, πολλοί από τους συνάδελφους αναφέρθηκαν στην ανεργία των νέων, αναφέρθηκαν επίσης και στις ε, μη καλές σχέσεις της παιδείας με ε, την οικονομία. Εσείς γνωρίζετε τα πράγματα Έχετε εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, ήσασταν υπεύθυνοι ανθρωπίνου δυναμικού σε μια πολύ μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, τώρα ασχολείστε με την πολιτική, έχοντας εν τω μεταξύ εργαστεί και σε μια μίκιο η οποία έχει σαν στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των σχολικών ιδρυμάτων. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε τις επαγγελματικές ικανότητες τις οποίες αποκτούν οι νέοι στα σχολεία με τις ανάγκες των μικρομεσαίων. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να καταρτήσουν οι ίδιες το προσωπικό τους. Οι καημένες όμως οι μικρομεσαίες δεν είναι σε θέση να κάνουν κάτι τέτοιο. Και αυτές είναι οι οποίες δημιουργούν κυρίως θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν σε ποιοτικό επίπεδο θα βοηθήσετε έτσι ώστε να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι ζούμε πλέον σε ψηφιακή περίοδο, σε ψηφιακή εποχή και γι' αυτό ε, οι υποδομές δημιουργούνται εύκολα και έχουν σαν στόχο να φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Ριμπάτσκα. Bardzo dziękuję. Z Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την κυρία Υπουργό. Έχω μόνο μία ερώτηση, διότι αυτά που θα ρωτήσω τα έχουν ήδη πει πολλοί ομιλητές Πώς τον προετοιμάσετε την διάσκεψη στην Αρμενία, την υπουργική διάσκεψη, κατά την άποψή σας, ε, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις επανεκκίνησης της διαδικασίας Μπολόνια. Ευχαριστώ συνάδελφοι, το λόγο έχει η κυρία Υπουργός. Αξιότιμα ε, μέλη. Μόλις έπαθε ένα ντεζαβού. Πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν εργαστεί στην παιδεία και στην κατάρτιση θα πρέπει να αισθάνθηκαν το ίδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραπαυτούμε στις δάφνες μας ο υπολογισμό των αποτελεσμάτων σε αυτό το τομέα δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε μεγάλη πρόκληση. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σα και τι ερωτήσει σα. Θα ήθελα να προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τι ερωτήσει και να τι απαντήσω με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ξεκινήσω με το γεγονό ότι εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε το εξής οι εργοδότες λένε ότι οι νέοι δεν ε, διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τις αγορές εργασίας. Η κυρία Αντενόφη ε, ανέφερε το ζήτημα αυτό. Και κατά τη συζήτηση με, τον Υπουργό Πολιτισμού, με την Υπουργό Πολιτισμού ανέφερε επίσης ότι ήταν απαραίτητο να σκεφτούμε πόσο σημαντική είναι η αναπτύξη της προσωπικότητας των νέων ατόμων. Τώρα αναφερόμενοι σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε την παιδεία με ευρύ πνεύμα, να έχουμε υπόψη μας την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ανταγωνιστικότητά μας θα εξαρτηθεί από τις δεξιότητες και τις ικανότητες των νέων μας. Από το πόσο μπορούν να αναπτύξουν την κρίση τους, να λαμβάνουν αποφάσεις και να είναι ανοιχτοί για νέες προκλήσεις. Η κυρία Ντενόλφη ανέφερε και κάτι άλλο. Το πρόγραμμα, το, το σχέδιο εγγύησης των νέων Είμαστε πεπισμένοι ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να, οπωσδήποτε να συνεχιστεί. Κατά την προεδρία μας θα κάνουμε μια αξιολόγηση του προγράμματος, θα δούμε τι ήταν επιτυχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και θα αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ διαφορών τομέων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του προγράμματος εγγύησης για τους νέους του Youth Guarantee Program. Η κυρία Σαμπίνα Φερχάινεν ανέφερε επίση ε, και το ζήτημα της ε, ανεργίας των νέων. Όπως έχω ήδη αναφέρει, η συνεργασία μεταξύ όλων των ε, επίπεδων παιδείας και της αγοράς εργασίας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όσοι από εσάς ε, έρθετε να επισκεφτείτε τη Λετωνία θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πώς οργανώνουμε τη συνεργασία μεταξύ του τομέα της παιδείας και της αγοράς εργασίας και πιστεύω ότι συμβαίνουμε ιδιαίτερη επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Τώρα για να απαντήσω την ερώτηση της κ. Βερχάινεν όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης ε, εκπαίδευσης θα ήθελα να τονίσω ότι μία από τις προτεραιότητες προεδρίας μας είναι να αναγνωρίζει την άτυπη εκπαίδευση όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Σπάρμπαλτ για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά του και για το ενδιαφέρον του εκφράζει στη διαδικασία της Μπολόνια. Πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν τη διαδικασία της Μπολόνια. Εγώ θα ήθελα να πω ότι προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε τους αρχικούς στόχους του προγράμματος το 1999. Τότε ο κύριος στόχος ήταν η ενίσχυση της κινητικότητας των νέων που είναι ουσιώδες, ε, ουσιώδης παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κατά τη διάσκεψη στο Γερεβάν, εμείς πρόκειται να ξαναδούμε τους αρχικούς στόχους και θα μελετήσουμε τα ζητήματα των πτυχίων, της αμοιβές αναγνώρισης τους αφενός, αφετέρου θα δώσουμε περισσότερη προσοχή στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Όπως ε, ανέφερε και ο κύριος Φέρ, η στάση προς τη διαδικασία της Μπολόνια είναι διαφορετική ανάλογα με το επίπεδο. Οπότε χρειαζόμαστε μια επανεκκίνηση της διαδικασίας αυτής. Η κυρία Γαμνή ότι είναι πολύ δύσκολο να διασφαλιστεί η ποιότητα και η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Είμαστε πεπισμένοι ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας θα δώσουμε προσοχή σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Ο κύριος Βέντ ε, αναφέρθηκε στον αθλητισμό. Ανέφερε την έννοια του διτού χαρακτήρα του αθλητισμού. Ναι, αναγνωρίζουμε αυτό τον ε, διτό χαρακτήρα του αθλητισμού. Αφενός είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να αγωνίζονται οι νέοι, να επιτυγχάνουν ε, πράγματα στον αθλητισμό κτλ. Αλλά αυτός είναι ένας από τους τρόπους για να αποκτήσουν οι νέοι τις απαραίτητες δεξιότητες και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και πιο ε, επιτυχείς στην εξέλιξή τους και στην, στα διαδρομία τους. Για το σχόλιο του κύριου Νέκος, ε, Θα ήθελα να συσχετίσω την ερώτησή του με το ζήτημα της αναγκαιότητας ευθυγράμμισης της επίσημης και της ανεπίσημης εκπαίδευσης. και της καλύτερης ευθυγράμμισης μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Αυτό αποτελεί μία από τις προτεραιότητες ε, της Προεδρίας μας. Προτεραιότητα για την Προεδρία μας είναι αυτή η ευθυγράμμιση, η μελέτη της. Σίγουρα θα συζητήσουμε και τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πληρέστατες οι απαντήσεις σας. Νομίζω ότι πίσω από όλες αυτές τις ερωτήσεις βρίσκεται το αίτημά μας προς την Λετωνική Προεδρία να προσπαθήσει ιδιαίτερα να προωθήσει τα πράγματα, ιδιαίτερα σε θέματα όπως η διαδικασία της Μπολόνια για να μπορέσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε με τον δικό μας τρόπο να ανοίξουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προς τον κόσμο, να είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους και να καταστήσουμε επίσης πολύ πιο προσβάσιμα τα πανεπιστήμια αυτά στους νέους πολίτες μας. Να ενταχθούν οι νέοι ε, στην διαδικασία αυτή κατάρτισης, να εμπλακούν οι νέοι ακόμα περισσότερο από ό,τι σήμερα μια περαιτέρω διεθνοποίηση του εκπαιδευτικού πανεπιστημιακού ευρωπαϊκού συστήματος. Και θα ζητήσουμε λοιπόν και από την υπηρεσία αυτή που έγραψε σε την έκθεση για την ανταγωνιστικότητα των πανεπιστημίων να μας δώσει την έκθεση σε περισσότερες γλώσσες για να δούμε ακριβώς σε ποιο βαθμό είναι προσβάσιμα τα πανεπιστημιακά αυτά δίκτυα στους Ευρωπαίους νέους ιδιαίτερα την εποχή της κρίσης. Και εκτιμούμε λοιπόν ιδιαιτέρως την προσπάθεια την οποία κάνατε έτσι ώστε να συνδεθεί ακόμα περισσότερο η επαγγελματική κατάρτιση με την κατάρτιση γενικότερα και με την επιχειρηματικότητα και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν βασική προτεραιότητα της Ιταλικής Προεδρίας άλλωστε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή, μας, παρέμβασή σας συγγνώμη, και για την παρουσία σας εδώ. Εύχομαι καλή δουλειά. Thank you very, very much and, hope to Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εύχομαι η συνεργασία μας στο επόμενο να αποδειχθεί πραγματικά καρποφόρος. Ε, cari colleghi, dear colleagues. Συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Σημαντικά σημεία και αυτά. Θα δώσω τώρα λοιπόν τον λόγο στη συνάδελφο Λιμπάτσκα. Θα μας παρουσιάσει η κυρία Λιμπάτσκα τη μία πρώτη ε, πρόταση αν θέλετε για την Πολόνια. Η πρώτη συνάντηση είχε γίνει το 12, ε, το 15 θα γίνει η δεύτερη διάσκεψη για τη διαδικασία αυτή στο Γερεβάν στην Αρμενία για τον Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Χώρο και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα ε, θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάποιες θέσεις σαν κοινοβούλιο σε, σωστό ε, χρονική, σε σωστή χρονική φάση. Η συγγήτρια θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της επόμενης συνάντησή μας την πρότασή της και η ψηφοφορία θα πρέπει να γίνει στις 24 Μαρτίου έτσι ώστε να φτάσουμε εγκαίρως στην Ολομέλεια του Απριλίου. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλύψουμε αυτό το ε, ουσιαστικό χρονοδιάγραμμα για την Επιτροπή μας. Κυρία Λιβάτσκα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω και την Λετονική Προεδρία. Η Λετονική Προεδρία έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά από ό,τι φαίνεται ήδη και θα πρέπει να περάσουμε τώρα στο θέμα της Μπολόνια. Να θυμίσω ότι η διαδικασία της Μπολόνια προσπαθεί από τη μία να δώσει απαντήσεις στην ανάγκη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση και από την άλλη να καλύψει τις ανάγκες ε, της πανεπιστημιακής παιδείας στον τομέα της καθολικής πληροφορίας και της ψηφιακής αγοράς. Η Μπολόνια καλείται να δώσει και απαντήσεις στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να αυξήσει τον ελκυστικό χαρακτήρα και την ανταγωνιστικότητα της ανώτατης ευρωπαϊκής εκπαίδευσης θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Οι Υπουργοί στην Πολόνια όρισαν τους βασικούς στόχους. Ο πρώτος από τους στόχους αυτούς ήταν να γίνει μια διάκριση των σπουδών σε δύο μεγάλες βαθμίδες. Στην διάσκεψη του Βερολίνου το 2003 καθορίστηκε και η τρίτη φάση σπουδών ταυτόχρονα υπήρξε και ε, μια προσπάθεια να καταστούν τα ευρωπαϊκά διπλώματα αναγνωρίσιμα παγκοσμίω. Ένα τρίτο θέμα το οποίο τέθηκε ήταν τα λεγόμενα credits, τα σημεία, οι βαθμοί δηλαδή, οι οποίοι μαρτυρούν τις γνώσεις τις οποίες έχει λάβει ο φοιτητής. Και το τελευταίο θέμα που συζητήθηκε ήταν η ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης ε, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συστημάτων ε, παραγωγής, αν θέλετε, επιστοποιητικών γνώσεων. Αυτές οι διαδικασίες καθορίστηκαν αλλά ταυτόχρονα ε, άλλαξαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Θυμίζω όμως ότι η διάσκεψη του Βερολίνου ήταν κρίσιμη γιατί ε, δημιούργησε το λεγόμενο τρίτο επίσης αμοιβαία των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών πτυχίων. Μια άλλη σημαντική διάσκεψη ήταν αυτή του 2005 που ασχολήθηκε με την έρευνα. Το 2011 έγινε μια άλλη μεγάλη συνάντηση στο Βουκουρέστι και εκεί καθορίστηκαν τρεις στόχοι για το 2015, ανύψωση της ποιότητας, αύξηση της απασχολησιμότητας των πτυχιούχων και αύξηση της κινητικότητας επίσης των πτυχιούχων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Βουκαρέστης συνεισέφερε από πλευράς του με μια εξαιρετική θα έλεγα έκθεση του ε, συναδέλφου Μπερλίνγκουερ. Φέτος το 2015 δηλαδή θα γίνει και η συνάντηση στο Γερεβάν και εμείς θα πρέπει να συνεισφέρουμε ε, στην διεξαγωγή της και γι' αυτό ακριβώς σήμερα ξεκινάμε μία πρώτη συζήτηση. Για να γίνει σωστά όμως η συζήτηση αυτή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε μέχρι τώρα το τι ήταν η διαδικασία της Μπολόνια και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας και ε, τους εξωτερικούς παράγοντες όπως την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη κτλ. Η διαδικασία αξιολόγησης της Μπολόνια δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν από τους υπέρ και τους κατά του συστήματος. Σαν παράδειγμα η διαδικασία 3 συν 1. Όλοι κάποιοι μάλλον λένε ότι ο φοιτητή μετά από τρία χρόνια μπορεί να μπει στην αγορά εργασίας. Κάποιοι άλλοι λένε μα πώς μπορεί κανείς να ολοκληρώσει σπουδές και να μάθει μια δουλειά σε τρία χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν ε, διαφορές και πράγματι σε κάποιους κλάδους δεν μπορεί κανείς σε τρία χρόνια να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ο κατάλογος λοιπόν των σπουδών που ακολουθούν τις παλαιές ε, ρυθμίσεις ε, παραμένει και το 90% όμως αυτών που ερωτήθησαν δεν συμφωνούν με τη διατήρηση των παλαιών συστημάτων. Ένα δεύτερο θέμα είναι το θέμα των HCTS, τα οποία θα πρέπει να αξιολογούν και να πιστοποιούν τις γνώσεις των, συνα... φοιτητών. Οι τελευταίες μελέτες μας δείχνουν, ιδιαίτερα σε σχέση με τις γερμανικές μελέτες, ότι μόνο το 50% των θεμάτων στα οποία κανείς εκπαιδεύεται στο εξωτερικό γίνονται αντικείμενο αναγνώρισης επίσημα από την χώρα καταβολής. Το πρόβλημα βρίσκεται ουσιαστικά στις νοοτροπίες του διδακτικού προσωπικού. Γιατί ε, ε, ο μοναδικός σωστός τρόπος για τους φοιτητές και τους καθηγητές των πανεπιστημίων είναι ο τρόπος που αυτοί επιλέγουν. Δεν μπορούμε έτσι να διασφαλίσουμε την σωστή κινητικότητα των φοιτητών. Ένα τρίτο θέμα. Τα εθνικά πλαίσια αναφοράς. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά γιατί ακριβώς δείχνουν το τι θα πρέπει να αποκτήσει σε επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων ο φοιτητής. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι τεχνητές οι ρυθμίσεις αυτές, καθόλου ε, πραγματιστικές. Οι συνάδελφοι μπορεί να έχουν τις απόψεις τους και μπορεί να συμφωνούν ή διαφωνούν. Πάντως, χθε οι Υπουργοί ανακοίνωσαν ότι θέλουν να ασχοληθούν κυρίως με τα θέματα της κινητικότητας και της διεθνοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι θα ασχοληθούν και με το αποτέλεσμα μιας ομάδας εργασίας που ασχολήθηκε με το θέμα της αυτόματης αναγνώρισης των τίτλων. Άλλοι θέλουν να ασχοληθούν με τα θέματα της λεγόμενης ανεπίσημης εκπαίδευσης, η άτυπης εκπαίδευσης. Άλλοι θέλουν να ασχοληθούν ειδικά και αποκλειστικά με το θέμα της ανώτατης εκπαίδευσης. Και λίγοι φοιτητές λέγουν ότι είναι ικανοποιημένοι από την παρούσα κατάσταση και ότι είναι λίγες οι δυνατότητες και οι ανάγκες βελτίωσης. Λοιπόν βλέπετε ότι όσες ερωτήσεις ε, θέτει κανείς άλλες τόσες απαντήσεις λαμβάνει. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε την κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Είναι μια κατάσταση σε ρευστότητα θα έλεγα, σε συνεχή εξέλιξη, υφίσταται τις πιέσεις της οικονομικής συγκυρίας, της δημογραφικής συγκυρίας, ε, επηρεάζεται από δηλώσεις Γιούνκερ για τις δυνατότητες ευρωπαϊκών επενδύσεων και θα πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα θέματα όπως το θέμα της πρόσβασης στις μελέτες. Έχει ενδιαφέρον το τι συμβαίνει στην Φιλανδία, ε, μια χώρα η οποία θέτει στόχους συγκεκριμένους ποσοτικά έτσι ώστε να ε, εγγυηθεί πλήρη πρόσβαση στην παιδεία για τις πιο εύθραυστες πλευρές της κοινωνίας. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε και για την εθνικοποίηση σε εισαγωγικά της διαδικασίας της Μπολόνια. Θα πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουμε παράδειγμα. Θα πρέπει να διδάξουμε στον διδάσκοντα ότι αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι η επιστήμη του, δεν είναι η αυλή του, αλλά η ουσία της εκπαίδευσης. Έτσι μόνο θα βοηθήσουμε τους φοιτητές. Λοιπόν, εγώ έκανα τώρα μόνο μια πολύ μικρή εισαγωγή. Θα μπορούσα να μιλήσω επί μακρόν και να περάσω σε λεπτομέρειες στην παρούσα φάση, αλλά δεν θα ήταν σωστό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να μου πείτε είναι κάποιες ιδέες τις οποίες έχετε για την πραγματική δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ανωτά της παιδείας. Λαμβάνοντας υπόψη πάντα την απαραίτητη πειθαρχία που πρέπει να χαρακτηρίζει τις επιστήμες. Την 22η Ιανουαρίου θα συναντηθώ με τους σκιώδεις εισηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων και την 29η θα συναντηθώ με τους εμπλεκομένους και συμμετέχοντες στην δημιουργία και τη θέση σε εφαρμογή της διαδικασίας αυτής της Μπολόνια. Τώρα χρονοδιάγραμμα, να λάβουμε υπόψη μας τον χρονισμό μετάφραση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για την κατάθεση των τροπολογιών. Σας προτείνω λοιπόν ε, να, καταθέσετε, να καταθέσουμε μάλλον όσο περισσότερες συμβιβαστικές τροπολογίες ε, γίνεται ήδη από τώρα να τις προετοιμάσουμε για να καλύψουμε το σύνολο των θέσεων της Επιτροπής Πολιτισμού και να μπορέσει η συνεισφορά μας στην διάσκεψη του Γερεβάν να είναι ουσιαστική. Συνεργαστείτε λοιπόν παρακαλώ μαζί μου και σας ευχαριστώ ήδη γι' αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη για την έλλειψη χρόνου αλλά το Γερεβάν είναι αύριο. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση, ήταν πολύ σαφής. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, στερινές προθεσμίες, αλλά θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε για τις χρήσιμες πληροφορίες που δώσατε. Δίνω τώρα το λόγο στην Πέτρα Κάμερβερτ που τον ζήτησε και θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους. Ναι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την Χριστίνα για αυτή την πρωτοβουλία η οποία είναι αναγκαία. Είναι ένα αμφίβολο ότι ο στόχος της Μπολόνια είναι σωστός. Ωστόσο είμαι πεπισμένη ότι σήμερα η διαδικασία αυτή της Μπολόνια χρειάζεται μεταρρύθμιση 15 χρόνια μετά από τη δημιουργία της, μετά από τη θέση ισχύ της. Δυστυχώς ε, πολλές ε, ελπίδες ε, μας δεν εκπληρώθηκαν. Ελπίζουμε λοιπόν να βρεθούν κάποιες λύσεις πριν από το σε μια εφημερίδα αναφέρθηκε ότι λείπουν ακόμα πολλά από τη διαδικασία της Μπολόνια. Λείπουν ε, δυνατότητες απασχόλησης ε, φοιτητών, ε, ότι λέγονται πολλά στη θεωρία αλλά στην πράξη γίνονται ελάχιστα και ότι οι φοιτητές δεν καταφέρνουν πάντα να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ε, μέσω της διαδικασίας αυτής. Πολύ συχνά συναντώ φοιτητέ και αυτό που ακούω διαρκώς ε, είναι τα ίδια παράπονα. Οι σπουδές είναι πολύ περιοριστικές, δεν μπορεί κανείς να σπουδάσει ό,τι θέλει. Ακόμη και όταν έχει θέσει κανείς στόχους με το Εράσμος, όπως για παράδειγμα, χάνει κανείς πολύ χρόνο. Χάνει σχεδόν ένα ή ενάμιση χρόνο. Διότι συχνά αυτά που σπουδάζει κάποιος στο ξένο πανεπιστήμιο δεν αναγνωρίζονται από το πανεπιστήμιο της χώρας του. Το πτυχίο δεν έχει ε, επαρκή αξία και ότι σε τελική ανάλυση με ένα απλό πτυχίο δεν είναι κανείς απαραίτητα απασχολήσιμος διότι οι επιχειρήσεις προτιμούν ε, ανθρώπους με μάστερ. Να σας παραθέσω κάποια λόγια ενός καθηγητή πανεπιστημίου. Δυστυχώς οι φοιτητές παραμένουν για περισσότερο χρόνο στα πανεπιστήμια, αποκτώντας όμως λιγότερες γνώσεις και δεξιότητες. Χρειαζόμαστε τώρα ε, προσόντα πιο καλά προσαρμοσμένα. Ναι, λοιπόν, ε, οι μελέτες που κάναμε στα πανεπιστήμια μας επέτρεψαν να, δούμε με πιο κρίσιμο βλέμμα την κατάσταση. Συμπεραίνουμε και πάλι ότι η έρευνα ήταν ο πρωταρχικός στόχος και σήμερα πρέπει να κάνουμε λίγο πίσω για να δούμε συνολικά αυτή τη διαδικασία της Μπολόνια η οποία σήμερα δεν επιτρέπει πολυτομεακό πρόγραμμα σπουδών όπως συνέβαινε στην εποχή μου. Ελπίζω λοιπόν ότι στη διάσκεψη του Γερβάν θα μπορέσει κάποιος να το πει καθαρά. Χρειαζόμαστε πραγματικά μεταρρύθμιση της διαδικασίας της Μπολόνια. Ναι, επίσης να πω ότι ναι, η απασχολησιμότητα ε, είναι κάτι προφανές, είναι απαραίτητο, αλλά δεν πρέπει να γίνεται με κάθε θυσία. Διότι αυτή τη στιγμή η θυσία που υφίστανται οι φοιτητές είναι υπερβολικά υψηλή. Ευχαριστούμε πολύ ο συνάδελφος ο κύριος Τσβέρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. να παρεμβώ ως χειώδης συζητητής ε, αυτής της έκθεσης. Η συγγήτρια κυρία είναι η κυρία Λεμπάτσκα. Την ευχαριστώ για το εξαιρετικό της έργο και τη συνεργασία της μαζί μας. Ελπίζω ότι η διάσκεψη του Γερεβάν θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και ότι η έκθεση αυτή θα αποτελέσει λειτουργικό στοιχείο για αυτή τη διάσκεψη. Προφανώς ε, η έκθεση πρέπει να είναι λίγο ευρύτερη, να καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να συμπεριλάβει και το Κοινοβούλιο σε αυτή τη φάση εξολόγησης της διαδικασίας της Μπολόνια. Ελπίζουμε ότι οι απόψεις μας ε, θα τεθούν σε εφαρμογή ε, Καλωσορίζουμε λοιπόν τη διάσκεψη του Ιερεβάν που θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Εμείς έχουμε θέσει ε, ένα, μια περιορισμένη προθεσμία για αυτή την αξιολόγηση της διαδικασίας της Μπολόνια. Εγώ συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες Πολλοί έχουν τεθεί στην μεταρρύθμιση της διαδικασίας της Μπολόνια για την τριτοβαθμία εκπαίδευση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά, τι πρέπει να κάνουμε, να μεταρρυθμίζουμε τη μεταρρύθμιση και να ξαναμεταρρυθμίσουμε τη μεταρρύθμιση της διαδικασία Μπολόνια. Ίσως ε, να χρειαζόμαστε ε, μια νέα όθηση ώστε να εξελιχθούν το συντομότερο οι αδυναμίες, οι λήψεις και να επιτευχθεί ο στόχος που είχαμε θέσει πριν από 10 χρόνια ότι δηλαδή η τριτοβαθμία εκπαίδευση της ε, Ευρώπης θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη με τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ασίας και με το σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλού να είναι πιο επικεντρωμένο, πιο αποτελεσματικό, υψηλότερης ποιότητας ε, και πιο συγκρίσιμο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα να προσανατολίζεται στα αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα να σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία. Μιλήσαμε για την τρίτη γενναία πανεπιστημίων. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει χάσει το μονοπόλιο των πανεπιστημίων που είχε πριν από χίλια χρόνια. Σήμερα Έχουμε ένα βιομηχανικού τύπου πανεπιστήμιο, το Humboldt, ε, το οποίο προχωρά με μεγάλη ταχύτητα. Θα χρειαστεί να αλλάξουμε τις δομές μας και την οτροπία μας για τα πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε πριν από 10 χρόνια. Κυρίως όμως ε, πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε το, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να είναι εφάμιλη. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με την τρέχουσα μεταρρύθμιση. Αλλά τώρα βέβαια το κλειδί δεν είναι η συγκρισιμότητα των σπουδών, αλλά η συγκρισιμότητα των ικανοτήτων των φοιτητών. Δηλαδή ο Έλληνας φοιτητής πρέπει να είναι το ίδιο ικανός και το ίδιο καταρτισμένος όσο και ο Γάλλος ή οποιοδήποτε άλλος. Υπό τη Σλοβενική Προεδρία το 2008 ξεκινήσαμε το, ξεκίνησε να λειτουργεί το, πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων που συνέβαλε σε κάτι και βάσει του οποίου θα πρέπει να αλλάξουν τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Και βάσει αυτού θα πρέπει στη συνέχεια να προσανατολίσουμε το σύστημα στην Ευρώπη, τα συστήματα παιδείας στην Ευρώπη ώστε να είναι συγκρίσιμα. Φυσικά εκκρεμούν πολλά ζητήματα ακόμα. Θεωρώ ότι η διαδικασία αξίζει τον κόπο και ε, τα θετικά αποτελέσματα είναι πιο πολλά από τα αρνητικά. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να επιταχύνουμε και να παγιώσουμε τη μεταρρύθμιση της Μπολόνια. Και εγώ θα παρευρεθώ στο Γερεβάν ε, και πιστεύω ότι αξίζει πολλά η έκθεση για την οποία συζητάμε. Ελπίζω κάθε χρόνο να έχουμε μια τέτοια αξιολόγηση. Δεν αποτελεί πίεση προς τα κρατημέλη, αλλά έκκληση ώστε να εξυγχρονίσουν την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση το ταχύτερο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις μετά και από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει τα τελευταία χρόνια για την μεταρρύθμιση του ε, διαδικασίας Μπολόνια. Το μπάτσελο να είναι πολύ σύντομο, να είναι δυνατόν να ε, γίνει και διαμονή στο εξωτερικό και ε, να προχωρήσει μετά. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να μην είναι μονάχα έξι εξάμηνα, όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρχει και στην Αλοδαπή. Και το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι η αναγνώριση της επιδόσεως. Αν θέλουμε να υπάρχει κινητικότητα, πρέπει και τα πανεπιστήμια να αναγνωρίζουν αμοιβαία την επίδοση στην ημεδαπή και την επίδοση στην Αλοδαπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαραγκάλ. Αφού άκουσα λοιπόν τις ε, παρεμβάσεις και της πρώτης Υπουργού και μετά και της ε, εισηγήτριάς μας για τη διαδικασία της Μπολόνια, εγώ είμαι θα έλεγα ο σκιώδης εισηγητής των Πρασίνων και έχω αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια σωστή δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα ακόμα και μέσα στο στενό χρονικό διάστημα. Τώρα, θα ήθελα ότι, να πω ότι γενικά αντιμετωπίζουμε θετικά την, τα 15 χρόνια λειτουργίας αν θέλετε αυτής της πρώτης εφαρμογής αυτού του συστήματος αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και μία κάποια θα έλεγα α, αναγνώριση ότι έχει υπάρξει μια καποια θα ελεγα αναγνωριση οτι πίστης στους τοπικούς, τους εθνικούς εταίρους, τους πανεπιστημιακούς που εφαρμόζουν το πρόγραμμα αυτό. Έχει αποχρωματιστεί λίγο το πρόγραμμα και έχει υπάρξει μια αίσθηση βολής γύρω από το θέμα αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να επιστρέψει η διαδικασία της Μπολόνια στην ουσιαστική της πραγματικότητα, στην αρχική της εικόνα, στα πλαίσια της αυθεντικής μεταρρυθμιστικής αυτής ε, ε, προσπάθειας. Όχι μόνο οικονομικού κόστους θα είναι η προσπάθεια αυτή, αλλά σε προσωπικό επίπεδο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο και σε θεσμικό επίπεδο. Δεν μπορεί κανείς να καταλήξει βέβαια σε τελικά συμπεράσματα και δεν γνωρίζω την πραγματικότητα που ισχύει σε όλες τις χώρες. Αλλά παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να καταλήξουμε όχι σε μια συνολική αντίληψη, αλλά να αναγνωρίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία και τον Μάιο θα έχουμε την δυνατότητα στο Γερεβάν να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική διάγνωση της κατάστασης και να προσπαθήσουμε να εργαστούμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να προωθήσουμε κάποιες κλίδες προτεραιότητας ε, για την ανάκαμψη της ουσίας αυτής της μεταρρύθμισης, να ξεκινήσει η λεγόμενη μεταρρύθμιση της μεταρρύθμισης δεν θέλω τώρα να παρουσιάσω λεπτομέρειες, να περάσω στο βάθος, αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς τους οποίους πρέπει να εμβαθύνουμε. Πρώτον, η πραγματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα μας επιτρέψει να έχουμε την συγκρισιμότητα την οποία έθεσε ο προλαλής σας. Διαφορές ανάμεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τους υπόλοιπους πανεπιστημιακούς χώρους όπως Κίνα, Ινδία, τα λοιπά. Θα πρέπει να αντικειμενικοποιήσουμε την κατάσταση αυτή για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε. Δεύτερον, να προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχει η ταύτιση του ρυθμού εφαρμογής της διαδικασίας της Μπολόνιας στις διάφορες χώρες και πόσον έχει επηρεαστεί η εφαρμογή αυτή ε, λόγω της μείωσης των δαπανών, λόγω της οικονομικής ε, ε, ε, στην χώρα μου όταν ε, λέμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε την Πολόνια και ταυτόχρονα μειώνουμε τις δημόσιες πιστώσεις για τα πανεπιστήμια και καταλήγουμε σε μια ηρωνική θα έλεγα αντιμετώπιση του προβλήματος. Και τρίτον, έχω την αίσθηση ότι τίθενται ορισμένες στόχοι από ορισμένους γενικού χαρακτήρα που δεν θα επιτρέψει μόνο τη συγκρισιμότητα αλλά και την βοήθεια για την περαιτέρω συστηματοποίηση του συστήματος της Βολόνια αλλά να υπάρξει μια μεγάλη ανύψωση των ποιοτικών στάνταρτς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσω της διαδικασίας της Μπολόνια ενός ευρωπαϊκού ποιοτικού σήματος για τα πανεπιστήμια. Ευχαριστούμε συνάδελφε Ραέν. Λοιπόν, Βεχίδεν, παρακαλώ να παραμείνετε σύντομοι γιατί πρέπει να τηρήσουμε τους χρόνους. Την αποδοχή στα ανώτατα σχολεία για αυτούς που έχουν τον μπάτσελορ από τα γερμανικά, από τις γερμανικές ανώτατες σχολές, γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη αντίσταση, υπήρχε τουλάχιστον στην αρχή, ειδικά ε, στις τεχνικές σπουδές, επέμεναν στο δικό τους πτυχίο. ενώ θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ελευθερία στην επίσκεψη και άλλων κύκλων μαθημάτων και ούτε καθεξής. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς διαμορφώνονται τα πράγματα αυτά. Το, η ανώτατη σχολή θα έχει ένα πρόγραμμα που ε, είναι άκαμπτο, που δεν μπορώ να παρακολουθήσω παρά μόνο μέσα στα πλαίσια του προβλεπόμενου έτους έχουν γίνει πολλά πράγματα εκεί που έχουν δυσκολέψει την διαδικασία ακόμη περισσότερο και σε ό,τι αφορά την αμοιβαία αναγνώριση. Σε κάποιους κύκλους σποδών, bachelor, μετράνε τα τάδε μαθήματα. Στο ε, πρόγραμμα για τον ίδιο κύκλο σπουδών σε, άλλη, σε άλλο πανεπιστήμιο βλέπουμε διαφορετικό συνδυασμό μαθημάτων για το ίδιο πτυχίο bachelor. Επομένω, δεν υπάρχει συγκρισιμότητα. Αν κάποιο έχει πάει ένα εξάμεινο σε άλλο δαπό πανεπιστήμιο, τα credit points που έχει δεν μπορούν να ενταχθούν πλέον στο αρχικό, στο πανεπιστήμιο της πατρίδας του. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Βεβαίω είναι επιθυμητή η ελευθερία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την άλλη μεριά, όμω χρειάζεται κάποια αποδοχή των ε, κύκλων μαθημάτων των άλλων πανεπιστήμιων. Πρέπει αυτό να μας προβληματίσει πώς θα κατορθώσουμε να επιτύχουμε κάποια συγκρισιμότητα των ε, ανωτάτων σπουδών. Αυτός ήταν και ένας από τους στόχους που υιοθετήθηκε το σύστημα Bachelor και Master και η διαδικασία της Μπολόνια να διευκολυνθεί πιο μακροπρόθεσμα η αναγνώριση των ε, πτυχίων. Έχω καμιά φορά την αίσθηση από πολλές ανώτατες σχολές, όχι μόνο ε, τις γερμανικές, ότι δεν υποστηρίζεται αυτό στην πράξη. Και εδώ πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια καλύτερη εξίσωση και να εξασφαλιστεί βεβαίω και η ποιότητα αλλά και η διάρθρωση. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου προηγουμένως, δεν μπορεί να είναι μόνο οι διαρροθετικές οι πρέπει να διασφαλίζεται και η ποιότητα. Βεβαίω η ευκαμψία, η ευελιξία υπάρχει. Υπάρχουν κύκλοι μαθημάτων bachelor, κάποτε το master είναι δύο ετών, άλλη φορά είναι τριών ετών. Αυτό το αποφασίζει το ΑΕΗ μόνο του και μέσα από τις δομές του. Υπάρχει λοιπόν τόσο μεγάλη ευελιξία και τόσο πολλές διαφορές που εν τέλει κάνουν δύσκολη τη συγκρισιμότητα. Ευχαριστώ. Μόργανο. Ευχαριστώ και εγώ να αναφερθώ σύντομα γιατί το θέμα αυτό χρειάζεται μέγιστη προσοχή. Το πρώτο όμως πρέπει να πω είναι το εξή. Μου φαίνεται ότι με όλα τα προβλήματα του ουσιαστικό ερώτημα είναι θέλουμε να προσπαθήσουμε να ε, κυβερνήσουμε, να, να ελέγξουμε, να διαχειριστούμε αυτό, την πολυπλοκο, το πολύπλοκο θέμα. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να βρούμε μια μέση οδό ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε κάποια συνεννόηση. Και φυσικά ο κόσμος δεν σταματά εκεί σε έναν κόσμο συνεχών αλλαγών ποτέ δεν επιτυγχάνεται οριστικό αποτέλεσμα. Δύο είναι τα προβλήματα. Η αυτονομία των ε, λυκείων ε, και η νομίμη ισχύς των πτυχίων. Διότι ξέρουμε ότι οι ρυθμίσεις διαφέρουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα και εκτός της Ευρώπης φυσικά. Νομίζω ότι διακρίνουμε την απέτηση που υπογραμμίστηκε και σήμερα με την παρουσία της Υπουργού που ήρθε να μας μιλήσει. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει για τη διακυβέρνηση της ε, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ε, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Μια τέτοια επιλογή στην Ευρώπη ε, Μα οδηγεί σε μια διαφορετική διαδρομή. Αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί κάποιες βάσεις δεδομένων των δυσκολιών που υπάρχουν. Πρέπει όμως να κάνουμε κάποια διάκριση. Όλα τα προγράμματα σπουδών ε, δεν χρειάζονται ε, το πρόγραμμα των τριών συν δύο ετών. Το τρία συν δύο αφορά πιο άλλου είδου σπουδέ και το μάστερ ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο και εδώ. Ορισμένα ε, σπουδέ σχετίζονται με άμεση είσοδο στην αγορά εργασία, άλλε ε, έχουν διαφορετική, διαφορετικό πρόγραμμα και διαφορετική διαδρομή. για ορισμένου τομείς είναι αδύνατον στο πανεπιστήμιο να παρακολουθεί το πανεπιστήμιο τι τεχνολογικέ εξελίξει. Συνεπώς ε, η Χριστίνα που υπογράμμισε προηγουμένως με μεγάλη ειλικρίνεια ε, το υποστηρίζω και εγώ. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε ξανά την υψηλή ποιότητα, την αποσχολησιμότητα όσα υπόθηκαν στο Βουκουρέστι, την έρευνα, ε, θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αναλύσουμε αυτή την εποχή. Κάτι θέλω να επιστήσω την προσοχή, κάτι στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Προσοχή γιατί σε ορισμένες χώρες Αφενός υπάρχουν επενδύσεις, αλλά η πανεπιστημιακή ζωή φαίνεται να είναι η τελική φάση της ζωής ενός ανθρώπου και δεν υπάρχουν δουλειές. Πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνεται αυτό. Και τέλος, όσον αφορά τις κατατάξεις των πανεπιστημίων, να θυμόμαστε ότι αυτές γίνονται βάσει υποκειμενικών κριτηρίων υπάρχουν πανεπιστήμια που κάνουν περισσότερη έρευνα και λιγότερη διδασκαλία. Άλλα πανεπιστήμια που κάνουν περισσότερη διδασκαλία ε, πλήττονται. Κάποιες χώρες προτιμούν τα μεν και κάποιες χώρες προτιμούν τα δε. Και δε, επίσης, ε, συνεπώς δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτές τις ταξινομήσεις, αυτές τις κατατάξεις των πανεπιστημίων και τις ικανότητες που προσφέρουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, Βέντα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ την κυρία Λουμπάτσκα για την παρουσίασή της. Ήταν μια πυκνή και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Υπάρχουν πολλά θέματα που άπτονται της ποιότητας της πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Μια στενότερη συνεργασία ανάμεσα τον επιχειρηματικό κόσμο και στον πανεπιστημιακό κόσμο να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Βλέπουμε την υπερπαραγωγή θα έλεγα μορφωμένων ανθρώπων σε ορισμένους τομείς όπου δεν χρειάζονται Ίσως η βιομηχανία και η οικονομία να μην είναι σε θέση να δώσει εγγυήσει για συγκεκριμένους αριθμούς πανεπιστημιακού τύπου απασχολούμενων, αλλά σίγουρα μπορεί να δώσει κατευθύνσεις. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τάισον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Συγγνώμη, Πρώτα θα πάρει το λόγο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέει στην εισηγήτρια ή πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένη για την πρωτοβουλία της Επιτροπής σας. Ξεκίνησε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία πριν τρία χρόνια με τον καθηγητή Μπερλίνγκουερ αν και η διαδικασία της Μπολόνια δεν είναι μια διαδικασία ενωσιακή, αλλά είναι κάτι στο οποίο υπολογίζουμε πολύ και πιστεύουμε ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο. Όπως είπαν και αρκετοί ομιλητές, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής για την Πολόνια. Πολλά έχουμε πετύχει, δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ διστακτικοί απέναντι στα επιτεύγματα ο, το σύστημα των τριών κύκλων έχει εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες, όχι με τον ίδιο πλήρη τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει υπάρξει πρόοδος. Τα σημεία, τα κρέντεξη CTAs καλύπτουν το 75% των μαθημάτων που διδάσκονται στα πανεπιστήμια και σχετικά με την αναγνώριση θα έλεγα ότι το 80% των φοιτητών του Εράσμους έχουν καλύψει τις ανάγκες τους. Υπάρχουν κενά αλλά έχουμε προχωρήσει. Υπάρχουν επίσης και θέματα ποιοτικής διασφάλισης. Έχει υπάρξει γενικά αρκετή πρόοδος. Όμως η εφαρμογή όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν ιδιαίτερος άνηση στις 47 χώρες που εμπλέκονται. Και είναι αλήθεια, μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και κουράζεται θα έλεγα, πρέπει να την ενισχύσουμε εκ νέου και νομίζω ότι θα το πετύχει η δική σας προσπάθεια. Ήδη έχει υπάρξει στο εσωτερικό της διαδικασίας της Μπολόνια μία επεξεργασία επανισχυροποίησης της εσωτερικής. Ίσως η διαδικασία να προσπάθησε να κάνει πάρα πολλά πράγματα ε, σε μικρό χρόνο και ίσως θα πρέπει να ε, ορίσουμε τις βασικές προτεραιότητες του 99 ξεχωρίζοντας αυτά που είναι αναγκαία για την διεθνοποίηση των πανεπιστημίων μας και την κινητικότητα των φοιτητών. Δεύτερον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε το τι πετύχαμε μέσω της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων. Όχι μόνο να πούμε το τι πρέπει να κάνουν οι χώρες μέλη, αλλά να τις βοηθήσουμε να τα κάνουν. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε και τις θέσεις των κρατών μελών εξ αρχής. Μιλάμε για χώρες από την Ισλανδία μέχρι το Καζακστάν. Η κατάστασή τους είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με τα συστήματα εκπαίδευσης. Απαιτείται λοιπόν διαφοροποιημένη αντίληψη που θα καλύψει τις ανησυχίες και τις προκλήσεις. Έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση από το 2012 και την διάσκεψη και ανακοίνωση του Βουκουρεστίου. Το πρώτο είναι η αύξηση της ανάγκης για διεπιστημονικότητα. Το είπαν αρκετά οι συνάδελφοι αυτό σήμερα. Οι πανεπιστημιακοί ομιλούν πολύ για την διεπιστημονικότητα, αλλά δεν κάνουν πάρα πολλά πράγματα και όταν κάνουν κάτι τότε το κάνουν στα πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και όχι στα μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια, όπου οι σχολές είναι απομονωμένες, είναι μεγάλες νήσοι λειτουργούσες αυτόνομα. Το θέμα επίσης της παγκοσμιοποίησης επηρεάζει την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε όχι μόνο τις κινήσεις στο εσωτερικό της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και <coughs> της ένταξης σε άλλες χώρες όπως η Λατινική Αμερική, η Βόρεια Αμερική και οι ανάγκες ε, ε, που αναγνωρίζουμε και στους χώρους αυτούς. Ε, προκλήσεις και προβλήματα από τη μείωση των δημοσίων ενισχύσεων. Αυτό είναι πρόβλημα για τα πανεπιστήμια σε πάρα πολλές χώρες που έχουν μειωθεί τα έσοδά τους από τις δημόσιες συνεισφορές κατά 20-25% λόγω της κρίσης. Η Μπολόνια δεν έχει δώσει απαντήσεις σε αυτό το πρόβλημα και πρέπει να το κάνει. Και τέλος, νομίζω ότι η ταχύτητα των εξελίξεων στον τομέα της πληροφορικής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της Μπολόνια. Η ψηφιοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης παρουσιάζει πολύ δυναμικό ιδιαίτερα στον τομέα της παγκοσμιοποίησης, αλλά και προκλήσεις και δυσκολίες σχετικές με τη διασφάλιση των μαθημάτων τα οποία γίνονται εκτός χώρας του Πανεπιστημίου ε, με φοιτητές που παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Πώς εμείς θα διασφαλίσουμε την ποιότητα αυτή, πώς θα ελέγξουμε και θα εξετάσουμε τους φοιτητές αυτούς καλύτερα. Είναι νέες εξελίξεις τις οποίες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε να βελτιωθούν μέσω της διαδικασίας της Πολόνια. Δεν είναι αργά για το Κοινοβούλιο να καταθέσει τις ιδέες του. Θα είναι ιδιαίτερα θετικό για τα πανεπιστήμια, για τους υπουργούς μάλλον πριν από το Γερεβάν, να ξεκαθαριστούν οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν στην ανωτάτη εκπαίδευση, πρέπει όμως να υπάρξουν κάποιες προτεραιότητες ε, στις οποίες να συγκεντρωθούν οι υπουργοί για τα επομενα τρια τρία-τέσσερα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ για τις προτάσεις ε, και τις εκτιμήσεις σας. Μας πιέζει πλέον ο χρόνος. Δίνω αμέσως το λόγο στη συνάδελφο κυρία Λίμπατσκα για τα συμπεράσματα ώστε να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους και όλες τους συναδέλφους ε, για τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους. Τρία είναι δίχως άλλο τα θέματα που ακούμε διαρκώς και διαρκώς, συνεχώς. Πρώτα απ' όλα η αναγνώριση των τίτλων σπουδών αλλά και η αναγνώριση των διαφόρων τμηματικών εκπαιδεύσεων προγραμμάτων που πιστοποιούνται με, τους, ε, με τις ακαδημαϊκές μονάδες, οι CTS. Ε, δεύτερον, είναι σημαντικό αυτό που είπε μια συνάδελφος ε, πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι η τριετία πρέπει να διαρκεί 6-7 εξάμηνα. Το σημαντικό είναι να οδηγεί σε έναν πρώτο τίτλο σπουδών, ο οποίος επιτρέπει στους πτυχιούχους να μπουν κατευθείαν στην αγορά εργασίας. Και μετά το τρίτο ζήτημα που ανέφερε η εκπρόσωπος Κομισιόν, η διεθνοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων σπουδών. Η διεθνοποίηση, ναι μεν, αλλά πραγματική δεν μπορεί να είναι απλά ένα πρόσχημα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η διεθνοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μια πραγματική ε, κινητικότητα των φοιτητών ε, ώστε να αξιοποιήσουν ολόκληρες τις δυνατότητες, όλες τις δυνατότητες ε, του, χώρου, του Ευρωπαϊκού Χώρου Σπουδών σε ακαδημαϊκό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επίσης χρειάζεται να συσχετίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε. Να ευχαριστήσω ξανά θερμά όλους τους συναδέλφους. Να ζητήσω συγγνώμη για τις ε, στενές προθεσμίες. Ε, ελπίζω να συνεργαστούμε στενά και επικοδομητικά. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως ακούσατε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τα μέλη και από την Κομισιόν ε, όπως είπε και ο Μπερλιγκουέρα πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση στη διαδικασία της Μπολόνια το είπαν και άλλοι εδώ είναι θεμελιώδου σημασία ε, να ακολουθήσουμε τις προτεραιότητες αλλά και τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει ενώπιση της στρατηγικής 2020 να αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των νέων που εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία. Έχουμε κάποια όρια όσον αφορά του πόρους βέβαια αλλά το να προβλέψουμε ότι πρέπει κάποια χρήματα του κοινωνικού ταμείου να χρηματοδοτούν και αυτή τη δυνατότητα συμμετοχής των νέων ε, είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει την προσοχή μας. Επίσης ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και θα το κάνετε, ξέρω, τη μελέτη που κάνετε για την προσπελασιμότητα ε, πρέπει να το υπενθυμίζουμε και να δώσουμε προσοχή στο δικαίωμα για, ευρωπαϊκές, για σπουδές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια ώστε να υπάρχει συμμετοχή. Δεν προσθέτω άλλα γιατί έχουμε ε, πλέον περάσει τους χρόνους, τους έχουμε εξελίσει τους χρόνους. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερη η έκθεσή σας, ε, να το ξέρετε και ε, ξέρουμε ότι οι προθεσμίες είναι πιεστικές, αλλά πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο. Να υπενθυμίσω επίσης ότι έχουμε και τη μελέτη για το ranking των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που θα μπορούσε να αξιοποιήσει και τις εκβάσεις, ε, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας, δηλαδή τι γίνεται στα θέματα ισότητας, διεθνοποίησης και προσβασιμότητας. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9. Τώρα έχουμε και κλεισμένο των θυρών την συνεδρία των συντονιστών να υπενθυμίσω ε, τις προθεσμίες ε, για την εκθεσία αυτή. Επόμενη συνάντηση 26 Φεβρουαρίου παρουσίαση της ε, έκθεσης της εισηγήτριας. Ευχαριστώ.